Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κήρυξω την έναρξη της ε, σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής μας ε, Βιομηχανίας. Θα ήθελα πρώτα να σας εξηγήσω το εξής. Ο εισηγητής κύριος Φερέιρα που έχει θέμα για τη γαλάζια οικονομία και είχε προγραμματιστεί για τις 9 κανονικά, ε, ζήτησε να αναβληθεί το θέμα του και δεν θα το συζητήσουμε. Και κατόπιν λοιπόν αιτήματος του εισηγήτου το ακύρωσε αυτό το θέμα, γι' αυτό και αρχίζουμε στις 9.30. Οπότε δεν θα συζητήσουμε σήμερα για την γαλάζια οικονομία, αλλά τέλη Μαΐου πάει. Και θα πάμε τώρα προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζομένη στα δεδομένα και ε, η συγκίτρια είναι η κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ. Εξού και αρχίσαμε στις 9.30. Και τώρα τι έχουμε Ο ημερησία διάταξη το 6, προϋπολογισμός 2016, και το 7 ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας κοινών μετάλλων. Αυτά τα δύο ε, τα έχουν αλλάξει σειρά μεταξύ τους, πρώτα το 7 και μετά το 6. Το 7 πριν το 6. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι γίνεται τώρα με τη γαλάζια οικονομία. Αυτό το να βάλουμε εντελώς, έχει το σημείο ολόκληρο μέχρι τέλη Μαΐου. Τι έγινε, υπάρχει πρόβλημα με τις μεταφράσεις, δεν ήταν ε, έτοιμες όλες και αυτό είναι ένα σοβαρός λόγος αναβολής, αν δεν έχουν μεταφραστεί τα έγγραφα σε όλες τις γλώσσες. Και το ζήτησε ο εισηγητής άλλωστε ο οποίος το έχει ελέγξει. Άλλα σχόλια για την ημερήσια διάταξη, όχι, από ό,τι βλέπω. Μπορεί να εγκριθεί λοιπόν έτσι, χωρίς άλλες αλλαγές, τα θέματα 5, 7 και 6 με αυτή τη σειρά. Ανακοινώσεις Προέδρου. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ε, Πολιτών για να απαγορευθούν τα πειράματα με ζώα έχει διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβολία Πολιτών έχει στόχο να καταργηθεί η ε, οδηγία για τη χρήση πειραματοζών για επιστημονικούς σκοπούς και ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει μια νέα πρόταση που να εξαιρεί τα πειράματα σε ζώα. Θα γίνει σχετική ακρόαση στις 11 Μαΐου 2015. Προσεχώς, δηλαδή τη Δευτέρα. 3 ε, με 6.30 το απόγευμα. Στην αίθουσα Γιάν 4Q2. Ήτρε συμμετέχει ω συνδεδεμένη επιτροπή. Καταλαβαίνετε ότι η αρμόδια επί της είναι η Επιτροπή Γεωργίας. Επόμενη ενημέρωση. Εχθές έλαβα μια γραπτή ερώτηση για γραπτή απάντηση προς το Συμβούλιο του κυρίου Τούρμες, για την οποία ακόμα δεν έχει λάβει ο ίδιος απόφαση εντός των προθεσμιών που προβλέπει το άρθρο 130 του κανονισμού μας. Και σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 130 εδάφιο 4, θα προτείνω να εγγραφεί το θέμα αυτό στην επόμενη ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας. Αυτά ως προς τις συνεδριάσεις μας και τις ημερήσεις διατάξεις. Um, uh, λοιπόν, επόμενο θέμα. Υπαρίθμ τρία έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 23ης και 24ης Μαρτίου 2015. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Ωραία, τα εγκρίναμε. Πάμε λοιπόν στο 5 προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα. Yeah, exactly. Mrs. Kappel. It was not before. Before it was not Madam Kappel. Sorry, it was my mistake because I said it's Mrs. Kappel. Was okay. Uh, towards uh, uh, thrive. Λοιπόν, λέμε προς μια εκμάθηση οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ. Εξέταση ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης. Ανταλλαγή απόψεων βάσει της προτάσεως ψηφίσματος. Αυτά είναι προς απάντηση της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα. Το σχέδιο ψηφίσματος ασχολείται με τα λεγόμενα big data ε, που έχουν πολύ μεγάλη ε, σημασία και δυνατότητες και οικονομικές και κοινωνικές. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε 45 λεπτά είχαμε προβλέψει για αυτό το θέμα. Και επίσης θα δώσουμε το λόγο για 5 λεπτά στην εισηγήτρια, 3 λεπτά στους συντονιστές και 2 λεπτά σε κάθε μέλος της ομάδας της Επιτροπής συγγνώμη, που θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Κάπελ έχει εισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Στις 6 Μαΐου έκανα το παρόν ψήφισμα που βασίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένας τομέας που έχει τεράστια σημασία αυτός για τη βιομηχανία, ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για ε, την κοινωνία των πολιτών και για τις νεοφύς επιχειρήσεις. Startup. Με υποστήριξαν πολλοί σκιώδεις και ευχαριστώ και τον Μίχαελ Μπόνι, τον Νάτο Σόρο, τον Ζόφσκι και τον Νταβίτ Μορέλη που ε, έκαναν και εκείνοι τις προτάσεις τους και μπορέσαμε να τις συμπεριλάβουμε το ψήφισμα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ενδιαφερομένους που τις περασμένες εβδομάδες είχαμε σειρά επαφών ε, πολλών ωρών και καταλήξαμε σε αυτή την πρόταση και πολλοί υπάλληλοι και συνεργάτες βοήθησαν τα μάλα. Η διαδικτύωση που προσφέρεται τώρα από τα big data ε, είναι τεράστια για συνεργασία σε διάφορους τομείς, σε διάφορους κλάδους, στην έρευνα, στην ανάπτυξη. Είναι πάρα πολλά και ποικίλα και τα πλεονεκτήματα και οι εφαρμογές από τη δημόσια ασφάλεια μέχρι το τραπεζικό σύστημα, τα ασφαλιστικά, κατασκευή ε, ε, διαφόρων εργαλειομηχανών, μηχανημάτων, αυτοκινήτων. Είναι η τέταρτη ε, βιομηχανική επανάσταση στη Γερμανία και στην Αυστρία 4.0, ε, η IPM, η Cisco, η Intel και άλλες τέτοιες εταιρείες πληροφορικής, ε, το ίντερνετ των αντικειμένων, Internet of Things, ο άνθρωπος και η μηχανή είναι σε πλήρη συνέργεια. Ε, και το θέμα είναι πώς θα βγάλουν λεφτά η Amazon ας πούμε με το cloud, η Netflix που είναι μια νέα εταιρεία ε, στην Αμερική πριν από τρία χρόνια δεν υπήρχε, 35% ήδη των στοιχείων χρησιμοποιεί και του τζίρου και ακόμα και η γερμανική σιδηρόδρομη. Είναι ένας τεράστιος κλάδος αυτό με τα δεδομένα ε, που ε, παρέχει ανεξάντλητες δυνατότητες αλλά στη Γερμανία και στην Ευρώπη σήμερα δεν έχουμε την τεχνολογία, της επενδύσεις, ε, το πλαίσιο και την προστασία των δεδομένων. Για να τα επιτύχουμε όλα αυτά Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και ε, υπάρχουν ε, πλεονεκτήματα ανταγωνιστικά πολύ μεγάλα. Οι αποφάσεις ε, θα οδηγήσουν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας τάξης του 5,6%. 1,9% αύξηση του ΑΕΠ και 234% ε, αύξηση ε, των θέσεων απασχόλησης μέχρι ε, το 2020 825.000 θέσεις εργασίας. Ανθεί ο κλάδος, ακμάζει, καλπάζει 40% το χρόνο, επταπλάσια μεγέθηση από τον κλάδο της πληροφορικής που έτσι κι αλλιώς ταχύτατα ε, εφαρμόζεται. Μόνο 1,7% όμως των εταιριών μας ε, τα χρησιμοποιούν και 41% δεν τα γνωρίζουν καν αυτά τα ε, big data. Το θέμα της προστασίας των δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, το ηλεκτρονικό έγκλημα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ευρυζωνικότητα, μια νέα υποδομή για cloud, όλα αυτά τα ζητούσαμε ε, και στην έκθεση της κυρίας Δελ το 2013 και το cloud computing. Για να εφαρμοστούν όλα αυτά μέχρι το 2020 χρειαζόμαστε 34 ε, δις για την ευρωζωνικότητα, 21 δις θα ε, έρθουν από το δημόσιο κομμέα. 92,4 δις χρειάζονται συνολικά και από τον ιδιωτικό τομέα ε, το Ταμείο Επενδύσεων και το, ε, τα διαρθωτικά ταμεία 21 δις, το είπα ήδη. BSM ε, ήταν η τεχνολογία 2G ε, τότε, τώρα έχουμε φτάσει περίπου στο 5G. Θα πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει ταχύτητα γιατί έχει μείνει πίσω. Ε, δεν έχουμε τεχνολογία, δεν έχουμε ε, χρήματα, δεν έχουμε υποδομές και αυτό είναι εμπόδιο για τις εταιρείες. Και η κατάρτιση υπολείπεται, δεν έχουμε ειδικού σε θέματα δεδομένων, το λέει αυτό και η έκθεση και θα πρέπει να βρεθούν απαντήσεις και να δοθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορώ να συνεχίσω, λέει ο ναι. ε, μπορείτε να φτάνετε στα συμπεράσματα. Ε, λοιπόν, ε, υπάρχουν διάφορα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει προφορικά. Ε, πώς θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ανταγωνιστική αγορά στα big data με καλές προϋποθέσεις για τον ανταγωνισμό ποιο είναι το πλαίσιο που θα δημιουργήσει βιώσιμο στο μέλλον ε, με στοχευμένες επενδύσεις και προστασία δεδομένων ε, για να ανταποκριθεί και στη δυναμική αυτή αγορά. Πώς θα αυξηθεί η συνειδητοποίηση ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να δραστηριοποιηθούν στα big data και να μπουν και οι ευρωπαϊκές εταιρείες σε αυτή την αγορά να ενισχυθούν για να μπορέσουν να αποδειχθούν ηγέτες. Πώς ε, θα δημιουργήσει προδιαγραφές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρότυπα, της προδιαγραφές ε, και ε, διατηρώντας και σεβόμενη την προστασία των δεδομένων ιδιωτικών και δημοσίων. Πώς λοιπόν θα βελτιωθούν τα δίκτυα, η ευρυζωνικότητα, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα για τις υπηρεσίες όπως είναι η κρυπτογράφηση και τα πρωτόκολλα και το ίδιο αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Το ξέρω ότι είναι εθνικό ζήτημα, ταυτόχρονα όμως θα είναι πάρα πολύ απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει κίνητρα και πρωτοβουλίες για να μπορούν τα κράτη-μέλη να παίρνουν δάνεια για να ε, τα βάζουν στα προγράμματα σπουδών. Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Και τώρα ο κύριος Μπόνια από το ε, ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μπάρμπαρα ε, Κάπολ ε, για την ε, ιδιαίτερα καλή εργασία της. Είναι πολλά τα θετικά σημεία τα οποία μπορούν να προκύψουν από την χρήση μεγάλων δεδομένων, αλλά βεβαίως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα καλό οικοσύστημα αυτών των μεγάλων ε, συστημάτων, αλλά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε διασύνδεση, δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για νέες τεχνολογίες όπως είναι το 4G, καθώς επίσης ε, και η δυνατότητα ε, διαμόρφωσης και χειρισμού των στοιχείων μέσα από την σωστή και ασφαλή αποθήκευση των στοιχείων αυτών. Δημιουργία πλατφορμών που θα πρέπει να γίνουν ε, με ουδέτερο τρόπο ανοιχτοί ε, στο σωστό ανταγωνισμό και στην ελεύθερη επιλογή. Θα πρέπει να αναπτυχθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία ε, στην τεχνολογία αυτή και κατά αυτή την έννοια τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας παίζουν σημαντικό ρόλο στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει οπωσδήποτε επίσης να υπάρξει τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν θα υποβάλω τροπολογία στην παράγραφο 15 έτσι ώστε να γίνει πιο σαφής αυτό. Η δεύτερη διάσταση είναι η διαθεσιμότητα. Η πρόσβαση στην ε, πηγή των ε, δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε πρόκειται για ειδικά, ιδιωτικά, ε, δημόσια ή εμπορικά δεδομένα. Θα πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες βάσει των οποίων μπορεί κανείς να μοιραστεί αυτά τα δεδομένα. Η προστασία των ιδιωτικών δεδομένων και η ασφάλεια είναι εκ των ουκάνευ ε, τα data sharing και η ιδιωτικότητα των στοιχείων θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, διασφαλιστούν έτσι ώστε να μπορέσει να ελευθερωθεί η αγορά και να αναπτυχθεί χωρίς πρόβλημα. Τρίτον, η διαλειτουργικότητα. Ε, για να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει μια εγκάρσια αποδοχή από όλες τις χώρες και από όλους τους παρόχους ε, και πρωταγωνιστές. Και αυτό θα πρέπει να γίνει βέβαια με συγκεκριμένους ε, διασυνοριακούς μηχανισμούς, σαφείς κανόνες που θα είναι εξίσου καθαροί και για την κοινωνία και για τους εμπορευόμενους οι υπηρεσίες και τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη η οποία ταυτόχρονα θα πρέπει ε, να διασφαλίσει την βιωσιμότητα όλων ε, αυτών που γνωρίζουν τις τεχνολογίες, που γνωρίζουν ε, την σημασία των μεγάλων δεδομένων και που έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν. Βεβαίως θα πρέπει, στα πλαίσια μιας, θα πρέπει αυτό να γίνει μέσα στα πλαίσια ενός συστήματος ανοιχτού και ανοιχτής διακυβέρνησης και ανοιχτών συνόρων. Ναι, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αργότερα, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σόλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ λίγο χρόνο χρειάζομαι έτσι ώστε να καλύψω ε, ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό Ευχαριστώ την συνάδελφο Κάπελ γιατί η εργασία της αποτελεί εξαιρετική βάση για να ξεκινήσει η συζήτηση. Όπως είπε και ο προλαλής σας, η οικονομία ε, η οποία θα έχει στη διάθεσή της τέτοια δεδομένα μεγάλης κλίμακος είναι ε, οικονομία η οποία μπορεί να δώσει νέα πνοή ε, σε όλες τις δραστηριότητες είτε είναι δραστηριότητες μεμονωμένων επιχειρήσεων είτε είναι δραστηριότητες έρευνας διοικητικές ή κυβερνητικές δραστηριότητες υπάρχουν λογισμικά τα οποία πλέον έχουν την δυνατότητα να αναλύσουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων που παλιότερα δεν μπορούσαμε καν να το φανταστούμε. Μπορούν να κάνουν συνδέσεις, συνθέσεις συγγνώμη, ε, μέσω λογισμικών τα οποία μπορούν ε, στην ουσία να ε, δημιουργήσουν και νέα γνώση, το λεγόμενο software machine learned. Επομένως δίνεται μία προστιθέμενη αξία, μία νέα αξία στα δεδομένα. Όταν μιλάμε όμως για δεδομένα μεγάλης κλίμακας, όσο περισσότερα είναι, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώσουν, θα αυξηθεί η αξία τους με γεωμετρική πρόοδο. Είναι ε, γι' αυτό λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να βάλουμε όλα τα στοιχεία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί. Εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε δύο δευτερόλεπτα να ασχοληθώ με ένα θέμα όχι μονάχα δημιουργούνται θετικές ευκαιρίες ε, για τις κυβερνήσεις, για την πολιτική, για την κοινωνία, για τις επιχειρήσεις, για τη διοίκηση, αλλά δημιουργεί, προκαλεί και κάποιες νέες απειλές. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε ε, συλλέγονται στοιχεία ε, ε, αναρρύθμιτα σε αριθμό τον οποίο δεν θα μπορούσαμε να τον είχαμε φανταστεί. Έχουμε, θα υπάρχουν στοιχεία για 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Θα ξέρουν ας πούμε τι κάνανε χτες και τι θα κάνουν σήμερα και ενδεχομένως θα είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τι θα κάνουν αύριο οι άνθρωποι αυτοί γιατί θα έχουμε στοιχεία για όλους. Ε, ε, τι νοσηδιοκτησία ιδιοκτησία θα είναι αυτά. Είναι ένα κοινό ε, κληροδότημα της ευρωπαϊκής κοινωνίας, άρα θα πρέπει να διατεθούν σε όλους έτσι ώστε να δημιουργήσουν αξία και όταν λέω να είναι διαθέσιμα σε όλους ενώ στην κοινωνία, στη διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Και κάτι άλλο. Ένα άλλο παράδειγμα, πολύ γνωστό το Facebook. Κατανοούμε το βαθμό συγκεκριμένης γνώσης που έχει καθένας για τον καθένα μας βάσει αυτού του Facebook. Ε, ε, τελειώνω ελπίζοντας ότι δεν ολοκληρώθηκε εδώ η συζήτηση για το Κοινοβούλιο. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δοσενόφσκι από την ΕΣΥΑΡ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, Θα ήθελα να πω ε, ότι θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις και πάρα πολύ χρήσιμες. Ε, πολλά από όσα προτείναμε έχουν συμπεριληφθεί στο ψήφισμα και δεν μπορώ παρά να το επενέσω να τις το αναγνωρίσω. Ε, κατάφερε πάρα πολύ καλά η συγγήτρια να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να αναπτυχθεί όλος αυτός ο κλάδος των δεδομένων μεγάλης κλίμακας, το big data. Το δείχνει αυτό η οικονομία. Είναι τεράστιος ο όγκος και είναι και τεράστια η πρόκληση από όλα αυτά τα δεδομένα. Είμαι πεπισμένος ότι σήμερα θα θέσουμε πολύ καλά θεμέλια για την προφορική αυτή ερώτηση και για το ψήφισμα. Η κυρία Κάπελ έχει κάνει εδώ καταπληκτική δουλειά και την ευχαριστώ και τη συγχαίρω. Θα ήθελα να τονίσω μερικά μία μόνο, τα οποία ανέφερε και η συγγήτρια. Η χρήση των δεδομένων μεγάλης κλίμακας συνδέεται στενά με τις ανάγκες, ε, τις επενδυτικές στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Χρειάζονται μεγαλύτερες υποδομές. Ε, αυτό μετεξελίσσει και προηγούμενα έγγραφα που είχαμε εκπονήσει εδώ στην Επιτροπή μας, έτσι ώστε αυτή η ε, πρόθεση και η ενίσχυση να πιάσει τόπο. Μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ καλά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρυζωνικό διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν δεν υπάρχουν αυτοί οι ενισχυμένοι διάβλοι επικοινωνίας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επεξεργαζόμαστε αυτά τα τεράστια ε, σε όγκο δεδομένα και σε κλίμακα για να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και στη συνέχεια. Ε, Θέλω να υποστηρίξω και τα super computing centers ε, που διαχειρίζονται δεδομένα μεγάλης κλίμακας και τεράστιο όγκο όπως είπαμε. Ε, χρειάζεται ειδική μεταχείριση και ειδικό χειρισμός γιατί είναι πολύ περίπλοκα όλα αυτά και τα προγράμματα τα πανευρωπαϊκά όπως είναι ο Κοπέρνικος ε, και κάποιες φωτογραφίσεις εναέριες αεροφωτογραφίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα χρησιμοποιήσουμε. Ε, είναι πολύτιμη δουλειά της εισηγήτριας, προσβλέπω στη συνεργασία μαζί της και στην επόμενη ε, συνάντηση που θα έχουμε σήμερα με τον Επίτροπο Άντσεπ θα μας βοηθήσει αυτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια και πάλι. Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και τα δεδομένα είναι μεγάλης κλίμακας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάλλας από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Κάπελ για τη δουλειά που έχει κάνει. Εν είδη γενικού σχολείου θα ήθελα, έλεγα ότι υποστηρίζω ε, τη θετική προσέγγιση της έκθεσης. Όντως συνιστά μια ε, μεγάλη ευκαιρία για την ευρωπαϊκή οικονομία και την κοινωνία το θέμα των δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Όμως ταυτόχρονα χρειάζονται επενδύσεις και όσοι εκπονούν την πολιτική θα πρέπει να περάσουν αυτό το θετικό μήνυμα στις επιχειρήσεις, ώστε να θεωρήσουν και εκείνες ότι αξίζει να επενδύσουν σε αυτά. Ε, η δημιουργία μιας ενίας αγοράς ε, ε, δεδομένων μεγάλης κλίμακας προς το υπολογιστικό νέφος και προς το διαδίκτυο των πραγμάτων. τι χρειαζόμαστε όμως γι' αυτό. Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο για να διευκρινιστούν ζητήματα που υπονομεύουν την εξέλιξη των δεδομένων μεγάλης κλίμακας και άρση των κολλημάτων για την ε, δημιουργία μιας μεγάλης αγοράς. Ε, μεταβιβασιμότητα παραδείγματος χάρη, φορητότητα, ιδιοκτησία των δεδομένων, διαφάνεια, τέτοιου είδους ζητήματα. Θα ήθελα να κάνω συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Στο άρθρο 10 μιλάμε για νέους αλγόριθμους. Δεν ξέρω εάν ισχύει αυτό ότι είναι ένα, είναι ένα μόνο εργαλείο ο αλγόριθμος. Ε, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς, όμως θα πρέπει εν αυτή περιπτώσει να αναφερθούμε και σε άλλα εργαλεία. Το ίδιο ισχύει για την ανάπτυξη ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος θα χρειαστεί να το διευκρινίσουμε διότι όταν μιλάμε για ίσους όρους ανταγωνισμού θα πρέπει να ξέρουμε σε έναν τομέα μεγάλης έντασης ως προς τα δεδομένα τι μπορεί να επηρεάσει τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. Επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα χρειαστούμε μια πλατφόρμα για την ε, ε, κοινή χρήση των δεδομένων. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει δεν να αναλάβει μια, έναν ηγετικό ρόλο. Στη ΣΥΠΑ ξέρω ότι η κυβέρνηση Ομπάμα ε, έκανε μια αναθεώρηση 90 ημερών ε, των δεδομένων μεγάλης κλίμακας για να κατανοηθεί το δυναμικό τους αλλά και οι προκλήσεις. Πρέπει να λειτουργήσει ως πρωτοπόρος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να θέσει το σωστό πλαίσιο για να αρχίσουμε να πραγματευόμαστε αυτό το ζήτημα. Χαίρομαι και προσβλέπω ε, με ανυπομονησία στη μελλοντική συνεργασία με την κυρία Κέπελ για αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Κάλλας, η κυρία Έρνστ από την κούρα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, είναι σαφές και θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι με το big data είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας ανάπτυξης που μπορώ να σκεφτώ τώρα ενώπιον μας. Και αν το παρατηρήσουμε, βλέπουμε ότι μας έχει πιάσει τώρα ο πυρετός της χρυσοθυρίας. Τρέχουμε όλοι για το Ελντοράδο. Το ξέρω ότι υπερβάλλω, το λέω συμβολικά. Μας έχει πιάσει, πιάσει τώρα μία φρενίτιδα δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι είναι τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας. Χρειάζεται έρευνα θεμελιώδης και στις μεταφορές. Και υπάρχει και μια δεοντολογία στην τεχνολογία και θα πρέπει να το συζητάμε και αυτό. Και η δεοντολογία της τεχνολογίας ε, είναι τι γίνεται με την ιδιωτική σφαίρα, την περίφημη ιδιωτικότητα γιατί εγώ θέλω εδώ να γίνω ε, η Κασάνδρα, ας πούμε, ή να σας πω ότι έχω επιφυλάξει. Υπάρχει ε, ένα ε, περιοδικό για κομπιούτερ που λέγεται Computer Woche και λέει ότι υπάρχει μια λύση για την χρήση του πελατολογίου και μπορεί ε, να μελετήσει τις προηγούμενες σχέσεις αλλά και τη μελλοντική συμπεριφορά ενός πελάτη. Κάνει ψυχογράφημα του πελάτη, ε, ε, τις παραμονές μιας απόφασης για αγορά ή για εμπορική συναλλαγή. Καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται όταν μιλάμε για big data, μεγάλης κλίμακας δεδομένα. Είναι μια συνολική πληροφόρηση και πώς εξασφαλίζεται η ε, αυτοδιάθεση, ας πούμε, η δυνατότητα του κάθε ανθρώπου να ορίζει τα προσωπικά του δεδομένα. Θα πρέπει αυτά τα θέματα να τα συζητήσουμε. Και υπό αυτή την έννοια ε, θέλω να σας πω ότι το σημείο 5, για παράδειγμα, ε, δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει. Τονίζει ότι η προστασία των δεδομένων και ευκαιρίες δεδομένων μεγάλης κλίμακας δεν αποκλείουν, λέει, το ένα τον άλλο. Τι θα πει αποκλείει. Θα πρέπει να συνάδουν το ένα με το άλλο. Τα προσωπικά δεδομένα έχουν να κάνουν με πρόσωπα. Εγώ αυτό εννοώ, ανθρώπου, θα πρέπει να προστατεύονται. Υπάρχει και νομοθεσία ευρωπαϊκή σχετικά. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτό το επίπεδο ε, πρέπει να γίνεται σεβαστό και το ευρωπαϊκό δίκτυο όπως και το εθνικό του καθενός. Γι' αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν χρειαζόμαστε απλώς ψήφισμα ε, με αυτό το θέμα για μια ακμάζουσα, ανθούσα, ξέρω εγώ, ε, αλλά να κάνουμε ένα ψήφισμα που να λέει big data και privacy, απολύτως το λέω ότι εκφράζω κάποιες αμφιβολίες και επιφυλάξεις και πάω κόντρα στο ρεύμα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια τεχνολογία, όσο ιδιοφυής και να είναι αυτή, ε, και να χρειάζεται νέα όθηση και υποδομές, όλα αυτά είναι σωστά, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε και ποιο ρόλο παίζει εδώ ο άνθρωπος, το πρόσωπο, για τα προσωπικά ζητήματα και δεδομένα έχουν σημασία. Ήδη από το design να μπαίνει η προστασία των προσωπικών δεδομένων από την αρχή του σχεδιασμού αυτής της προσπάθειας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ταμπουράνα από το e Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο εισηγητή μα δυστυχώ είναι αυτή τη στιγμή σε άλλη επιτροπή. Μου ζήτησε να ευχαριστήσω την κυρία Κάπελ εξ ονόματό του για την ε, ε, συνεργασία που είχαν μέχρι τώρα. Και εδώ μεταφέρω και τα δικά του λόγα. Είμαστε απολύτω πεπισμένοι ότι θα πρέπει να δραχθεί η ευκαιρία ε, τη σωστή, ισορροπημένη και μακρόθωρη χρήση των δεδομένων δεδομένων και των δυνατοτήτων που η χρήση των δεδομένων αυτών μας δίνει. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή και επομένως ε, θα πρέπει να υπογραμμιστεί το σημείο αυτό από την, ε, ε, από την προφορική ερώτηση. Το θέμα της εσωτερικής αγοράς είναι πάρα πολύ σημαντικό και επομένως είναι απολύτως συνδεδεμένη η εργασία μας με το θέμα της εσωτερικής αγοράς. Εκεί θα πρέπει να ρίξουμε την ιδιαίτερη προσοχή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Άλλοι συνάδελφοι από πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούν πολιτικές ομάδες δεν υπάρχουν, οπότε περνάμε στα μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ ε, για τις προτάσεις ε, είναι πολλές οι ευκαιρίες που συνδέονται με τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας. Πολύ ωραία τα λέει το ψήφισμα και εστιάζει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για μένα είναι και σωστό αυτό και σημαντικό. Όσο και αν μας έχει πιάσει ενθουσιασμός όμως, θα πρέπει να δούμε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτό. Το είπε προηγουμένως η συνάδελφος, η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ε, και ε, εγώ θέλω να αφαιρθώ στην προστασία των εργαζομένων. Υπάρχει μια τάση ε, κυριαρχίας στην αγορά, ε, στα big data και στοιχεία ε, που δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα μπορούν να παρακολουθούν τις επιδόσεις αλλά και τη συμπεριφορά των εργαζομένων παρακαλώ και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εδώ. Η διαφάνεια της προέλευσης των προσωπικών δεδομένων είναι δεδομένη και αυτή και σε ποιον ανήκουν ε, τα δεδομένα και ποιος μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Στο σημείο 13 θεωρούμε ότι δεν είναι πολύ υψηλέ οι τιμές για τις ευρεσιτεχνίες γιατί έτσι ε, δημιουργούνται και κίνητρα για να επενδύει κανείς την έρευνα και την ανάπτυξη. Υπάρχουν και άλλες εταιρείε μη ευρωπαϊκές που έχουν ε, συμφέρον να μειωθούν οι τιμές. Και έχω μια ερώτηση ε, για αυτά που λέτε για τις θέσεις εργασίας. Στην παράγραφο 2 αναφέρονται κάποια στοιχεία ε, που συνδέονται με μία μόνο μελέτη ε, της Μεγάλης Βρετανίας του 2013 και αφορά το διάστημα μέχρι το 2018. Αυτή είναι η πηγή σας ή έχετε και άλλη πηγή, γιατί μόνο εκεί τα έχω βρει μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Ντεκαστήγιο. Ευχαριστώ πρόεδρε θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια γιατί είναι πάρα πολύ καλή η δουλειά της και παρουσιάζει και τις ευκαιρίες που έχουν τα big data. Ε, αναφέρεται στις ε, βασικές προκλήσεις, έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία, υποδομές, ε, όλα αυτά τα λέει πάρα πολύ ωραία. Τις ηλεκτρονικές δεξιότητες που χρειάζεται ο καθένας να έχει για να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες κτλ. Εγώ θέλω να προσθέσω μόνο μία διάσταση που υπονοεί το ψήφισμα, αλλά θα πρέπει να την πούμε πιο ξεκάθαρα. Και αυτό είναι η ευκαιρία που αποτελεί για την ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία το να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί παγκοσμίω. Όχι μόνο τι σημαίνει αυτό για μας θέμενη αξία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Όλα αυτά τα στοιχεία που συνδέονται καλώς, όπως η δημιουργία ε, ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη, αλλά πώς τοποθετείται η Ευρώπη ως οικονομία και ως ανταγωνιστικός ε, παράγων παγκοσμίω. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια, δεν ξέρω, ε, με σδίτ ενδεχομένως, για να εκπονήσουμε διάφορα πρότυπα για τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας, για να μπορέσει η Ευρώπη να έχει αυτή τη θέση που έχει. Που είχε ε, στις προδιαγραφές τα κινητά τηλέφωνα στη δεκαετία του 90. Και σήμερα προτείνει πολύ ευφυώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάπτυξη, γιατί ακόμα σε αυτή τη φάση είμαστε έρευνας και ανάπτυξης της τεχνολογίας πέμπτης γενεάς. 5G όπου οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρωτοστατούν. Υπάρχει αυτή η διάσταση διεθνούς ανταγωνιστικότητας και παγκόσμιου ανταγωνισμού από τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας και ανάγκη να δούμε ποια είναι τα πρότυπα ε, παγκοσμίω πάντα. Και εγώ θα κάνω κάποια τροπολογία σχετικά. Και πάλι συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ε, Πολύ σας ευχαριστούμε. Ζωρίνιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω και την εισηγήτρια και την, τους συνεργάτες της για την έκθεση που εκπώνησαν. Είναι εξαιρετικά επίκαιρο το ζήτημα, διότι έγινε πριν από την παρουσίαση ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το ενιαίο ψηφιακό ε, πλαίσιο με ε, το 5G έχουμε μία νέα ευκαιρία και δεν μπορούμε να χάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας σε παγκόσμια κλίμακα. Όμως ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι η οικονομία μας, ε, η οικονομία, συγγνώμη, θα πρέπει να εξυπηρετεί τους ανθρώπους και όχι το αντίθετο. Είναι μια ανθρωπιστική αρχή που πάντοτε ε, πρεσβεύουμε. Χρειαζόμαστε επίσης διαλειτουργικότητα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Πέρα από τις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να είμαστε γενικότερα διαλειτουργικοί. Οι θα πρέπει οι ίδιοι να είναι και ασφαλείς και διαλειτουργικοί. Μόνο έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα έρισμα κρατεό για αυτήν την ε, ενιαία ψηφιακή οικονομία. Κλείνοντας, ε, θα έλεγα ότι θα πρέπει οι ανθρώπινοι πόροι των μικρών επιχειρήσεων να είναι οι πρώτοι που θα υποφεληθούν από αυτήν την επανάσταση. Πέρα από τις νέες τεχνολογίες και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην αιχμή των νέων τεχνολογιών, γιατί εκείνες μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν, θα πρέπει οι, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη συνέχεια οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετάσχουν επίσης σε αυτήν την νέα επανάσταση. Την επανάσταση που κατά τη γνώμη μου θα έχει θετικά αποτελέσματα και για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε κύριε Ζωρίνιο. Κυρία Κούπουλα, Κούμπουλα Νάτρη, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω. Είναι εξαιρετική η έκθεση και πολύ θετική η προσέγγιση που υιοθετήσατε. Θα έχουμε καταπληκτικές ευκαιρίες νέες δυνατότητες εάν τηρηθούν και οι απαιτούμενες ε, ε, δικλείδες ασφαλείες μέσα σε αυτή τη νέα οικονομία. Για την ε, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, για την αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία της ψηφιοποίησης των δεδομένων. Για τις φορολογικές δηλώσεις, παραδείγματος χάρη, στη Φινλανδία οι πολίτες δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα για τις φορολογικές τους δηλώσεις. Είναι προσυμπληρωμένα τα έντυπα και επεμβαίνουν μόνο αν έχουν ε, κάποια διόρθωση να κάνουν. πώς θα επιβιώσει και θα εξελιχθεί η Ευρώπη σε αυτήν την παγκοσμιοποιημένη ψηφιακή οικονομία. Όταν στην Ευρώπη πάσχουμε από τις διαφορετικές γλώσσες που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Επίσης, νομίζω θα πρέπει το σημείο 5 να διορθωθεί. Σας ευχαριστούμε, ο κύριος Μαραγκάρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, όπως όλοι οι ομιλητές σχεδόν, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ την εισηγήτρια και να την ευχαριστήσω για το έργο της. Συμφωνώ και με τον κύριο Ζωρίνια. Άκουσα τι είπε η εισηγήτρια και η Λυπή, διάβασα και το ψήφισμα. Βεβαίως θα ήταν πάρα πολύ θετικό να συνδέσουμε τη συζήτηση αυτή με τη συζήτηση για τη διαλειτουργικότητα και τις δημόσιες επενδύσεις στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και θα πρέπει να είμαστε και συνδεδεμένοι και συντονισμένοι με αυτά. Υπάρχουν δύο θέματα για, το, ερωτήσεις που έχω. Μία για το δημοκρατικό έλεγχο και τη ρύθμιση και το άλλο έχει να κάνει με τη τεχνολογία. Η προστασία των δεδομένων είναι πολύ σημαντική, αλλά και τα θέματα ρύθμισης, ανταγωνισμού, πρόσβασης, δυνατότητας, ε, πρόσβαση στην αγορά, στη ζήτηση και στην προσφορά. Εδώ νομίζω υπάρχει ένας κίνδυνος ανισοτήτων, δηλαδή αυτός που έχει τα big data είναι σε πλέον εκτική θέση, έχει όλες αυτές τις τεχνολογικές δυνατότητες, ευρυζωνικότητα, cloud computing κτλ. Ε, και θα πρέπει να προωθηθεί και η συλλογική χρήση ε, όλων αυτών των φανταστικών δυνατοτήτων με καλύτερη οργάνωση και των δημοσίων υπηρεσιών και υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση για ιδιωτική χρήση η οποία θα πρέπει να θωρακιστεί με προστασία και ασφάλεια. Υπάρχει και ένα θέμα τεχνολογικό που έχει να κάνει ε, με αυτό που είπε η κυρία Έρνστ, δημοκρατικός έλεγχος. Θα πρέπει οι πολίτες να ξέρουν ποιες είναι οι δυνατότητες, ποια είναι τα όρια, τι μπορούν να ε, ελπίζουν, τι κινδύνους μπορούν να διατρέχουν. Συνήθως συνδέουμε τα big data με ε, τους μεγάλους ομίλους, με τα big corporations. Αλλά να μην περάσουμε από το big data στο big brother. Αυτό είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος και θέλει προσοχή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Το διαπιστώνετε όλοι και τώρα ήρθε η ώρα για την Επιτροπή. Κύριε Λογιόλα Ντεσόλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Δεν είμαι σε θέση να κάνω ιδιαίτερα σχόλια όσον αφορά τα big data δεδομένα μεγάλης κλίμακας. Να σας πω πάντως ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει τη στρατηγική της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς, της οποίας σημαντικό στοιχείο είναι τα δεδομένα μεγάλης κλίμακος. Επομένως θα, λάβετε, θα δείτε όλες τις ιδέες που έχουμε και, όσον, και όλες τις δράσεις που ε, προϊονίζονται για τον τρίτο ε, πυλώνα. Ε, αυτά ήθελα να σας πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το περιμέναμε. Ως απάντηση της Κομισιόν. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας και θα ζητήσω από την κυρία Κάπολη τώρα να δευτερολογήσει προσπαθώντας να κάνει μια σύνοψη της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Το τελευταίο αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Θα έρθει και ο κύριος Άνσιπ στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσει τη νέα στρατηγική και δεν θα σας εκπλήξει ε, που το συνδέω και με την έκθεσή μου. Για να απαντήσω σε κάτι που ρώτησε η κυρία Βένερ στο σημείο 2 δεν αναφέρεται σε στοιχεία από το Ενωμένο Βασίλειο, αλλά στοιχεία που μας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως ήμασταν σε επαφή με την Επιτροπή. Το Big Data, όπως είπε και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, στοιχείο και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάζεται σήμερα. Και από πλευράς Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό να επιληφθούμε κι εμείς. Ε, και ήδη προεξοφλούμε διάφορα θέματα που θα παρουσιάσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νομικό πλαίσιο κτλ. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στην παράγραφο 5, στην οποία αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι, για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων. Αυτό ήταν ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για μένα και κομβικό και μόνο ακροθυγώς το εξετάζουμε, διότι θεωρούμε ότι είναι θέμα που χρειάζεται ξεχωριστό ψήφισμα και ξεπερνάει τα πλαίσια της Επιτροπής μας, Ήτρε, κατά πολύ. Βέβαια, σε όλη μας τη δράση στο κέντρο είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ούτε η βιομηχανία ούτε η οικονομία. Γι' αυτό η προστασία και ασφάλεια των δεδομένων και η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στα big data χρειάζεται και αξίζει ένα ξεχωριστό ψήφισμα και πολλές συζητήσεις και πολλές διαβουλεύσεις. Θα προσπαθήσω εγώ να το κάνω και με χαρά με τους σκιώδεις ηγητές τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Ίσως η παράγραφος 5 χρειάζεται καλύτερη διατύπωση για να το πούμε πιο ξεκάθαρα και να αναφέρουμε ότι θα υπάρξει και νέο ψήφισμα μόνο για αυτό το θέμα. Προσβλέπω στη συνεργασία τις επόμενες εβδομάδες σήμερα από άλλους ομιλητές αλλά κυρίως από τους σκιώδεις άκουσα ε, πολλά χρήσιμα. Τα σημείωσα ως ιδέες με χαρά να τα εντάξουμε στο ψήφισμά μας. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών κατάφερε να ε, παραταθεί. Δεν είναι η 12η Μαΐου πλέον, έχουμε μερικές μέρες παραπάνω. Θα κάνω και εγώ τροπολογίες, έχουμε χρόνο ακόμα. Ε, δεν μας έφτανε ο χώρος που είχαμε, πέντε σελίδες είναι πολύ λίγο για ένα τέτοιο τεράστιο θέμα. Λοιπόν, 15 Ιουνίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας το ψήφισμα και το Σεπτέμβριο αναμένεται να πάει στην Ολομέλεια. Και αφού ακούσουμε τον Επίτροπο ε, σήμερα, σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να συμπεριλάβουμε και άλλα στοιχεία. Προσβλέπω και χαίρομαι για τη συνεργασία με τους ε, σκιώδης και εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Κάπελ, ευχαριστώ Μπάρμπαρα για τις παρατηρήσεις σου. και για το συμπεράσματα που έβαλες. Προετοιμάζουμε λοιπόν προφορικό ερώτημα και ψήφισμα. Το αποφάσισαν οι συντονιστές της Επιτροπής μας να αναλάβουν το σημείο αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό ε, θέμα. Και επομένως ανταποκρίθηκε θετικά η Επιτροπή Ήτρε. Όπως και εσείς είπατε κυρία Κάπαλα, όσον αφορά τις τροπολογίες, η προθεσμία έχει οριστεί για την 12η Μαΐου του 2015, η ψήφος στην Ήτρε ενδεχομένως 16 Ιουνίου. Ψήφος στην Ολομέλεια ενδεχομένως τον Σεπτέμβριο μετά τις διακοπές. Προχωράμε τώρα στο επόμενο σημείο. Είναι η αποστολή στο Μπέρεκ. Regulators Πρόκειται για το σώμα των ρυθμιστών, ε, το, ρυθμιστών της ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ρυθμιστές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λέει ο Πρόεδρος, Μπέρεκ. Ε, which Λοιπόν, για τα θέματα αυτά είναι υπεύθυνη η ΙΤΡΕ. Γιατί εμείς ε, είμαστε υπεύθυνοι για τις τηλεπικοινωνίες και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Επομένως, στο Μπέρεκ και στο, στην υπηρεσία Μπέρεκ στην Ρήγα έγινε αυτή η επίσκεψη. Ε, συναντήσαμε τους υπευθύνους εκεί και πρέπει να σας πω ότι η αντιπροσωπεία της Ήτρε, η συνάδελφή ήταν ο κ. από το ΕΛΚΑ, και η Μισελ Ράι, ο Μισελ Ράιμουνα από τους Πράσινους. Ε, και από τους σοσιαλιστές η Κωνσταντσε Κρέλερ. Και ο Κάρινς ήταν παρόν, εκπροσωπούσε φυσικά τη Λετωνική Προεδρία εκεί. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν σε ανέφερα. Ο Γκούναρ Χέκμαρκ θα μπορούσε να κάνει ένα debriefing. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου ζητήσατε οτιδήποτε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να τονίσω πως είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Βιομηχανίας, ε, το ΠΕΡΕΚ. Έχω την κυρία Τελκαστήλιο εδώ και μπορεί να με διορθώσει. Θα έλεγα ότι παίξατε καταλητικό ρόλο πριν από λίγα χρόνια για να συγκροτηθεί ο φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τον Μπερέκ. Πρώτη φορά που πήγα στη Ρήγα έπρεπε να περάσω από τα φυλάκια της ε, ΚΑΓΕΜΠΕ. Αλλά τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το αντίθετο ισχύει τώρα. Πήγα σε μια από τις πρωτεύουσες Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν οργανισμό που βρίσκεται εκεί. Μεγάλη καμπή. Πολύ χάρηκα, πολύ περισσότερο από την πρώτη φορά που πήγα στη Ρήγα. Υπέροχη αυτή η πόλη. κύριος Μπαρός ε, είναι ο πρόεδρος για το 2015 και ο αντιπρόεδρος, ε, ο Δόκτωρ Βίλεμ Άισφέλερ, θα αναλάβει πρόεδρος για το 2016. Ο Λάτζιν Γκέντσι είναι ο μάνατζερ ε, για τα διοικητικά ζητήματα στον Μπέρεκ. Υπήρχαν και βουλευτές υπό τον κύριο Έντβαν Στίλτον. Συζητήσαμε για το ρόλο της λειτουργίας του Μπερέκ δεν έχει νομική προσωπικότητα. Ο οργανισμός ε, ανανεώνεται το προσωπικό πάρα πολύ συχνά. Νομίζω ότι για τεχνολογικά στήματα αυτό είναι πολύ θετικό. Και συζητήσαμε το θέμα του roaming, ε, της περιαγωγής. δύσκολα μπορούμε να ξεφορτωθούμε το κόστος περιεγωγής όσο οι υπάροχοι ε, παρόλα αυτά πρέπει να πληρώνουν κάποιο κόστος. Συζητήσαμε λοιπόν εκτενώς για το πώς θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Η κυρία Ντελκαστήγια όπως και άλλοι στην Επιτροπή ασχολούνται με αυτό το ζήτημα τακτικά. Ε, ο Μπέρεκ αυτό μας είπε ότι πρέπει να καλύψουμε με κάποιο τρόπο το κόστος ε, που ε, βαρύνει τους παρόχους για να βρεθεί μια λύση. Μιλήσαμε για την ουδετερότητα του δικτύου επίσης. Οι εθνικές διευθυντικέ αρχές έχουν εξαιρετικά αποκλίνουσες απόψει. και ο Μπέρεκ δεν έχει μια νέα γραμμή. ο Μπέρεκ, ε, θα έβγαζα εγώ ένα προσωπικό συμπέρασμα, ε, διαφέρει ως προς τη δομή του σε σχέση με τα, αυτά που είχε προγραμματίσει αρχικά ε, το Κοινοβούλιο. Είναι το αθρηστικό αποτέλεσμα εθνικών ρυθμιστικών φορέων. Δεν ξέρω αν η κυρία Καλίσκα συμφωνεί, αλλά... Κυρία Κρέλιο, Κάριν συμφωνούν, μπορούν να μας πούνε τι πιστεύουν. Ε, εγώ πιστεύω και το είπα πάντως ότι εξυπηρετούνται μόνο τα συμφέροντα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ε, παρά το γενικό, το δημόσιο συμφέρον. Ε, είναι δύσκολο βέβαιως να οριστεί αυτό. Όμως τα φεουδά τους υπερασπίζονται και θεμητό. Τα κατοχερωμένα πρέπει να τα προφυλάσσουμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ένα ευρύτερο όραμα. Το συζητήσαμε λοιπόν επί μακρόν και μου έκανε εντύπωση διότι διακεκριμένα μέλη των Εθνικών Εθνιστικών Φορέων και του Μπέρεκ μας είπαν ότι Όλα αυτά τα προβλήματα μπορούμε να τα ρυθμίσουμε στα πλαίσια εθνικών ρυθμιστικών ε, διατάξεων. Δεν είμαι ε, ακρεφνής φεντεραλιστής ε, προσωπικά, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι μια κοινή προοπτική για τη χρήση του φάσματος, παραδείγματος χάρη, για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών δικτύων θα μπορούσαμε να έχουμε. Και γιατί σας το λέω αυτό, διότι... Ένα μεγάλο τμήμα της αξιολόγησης που κάνει ο Μπέρεκ σχετίζεται και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι με το να εξασφαλίσει ότι δεδομένων των συγκυριών και των προϋποθέσεων που έχουν προσδιοριστεί προσπαθεί να έχει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Ωραία, καλό, αλλά πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή την υποδομή. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Εγώ προσωπικά Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή δυναμική για να άρουμε αυτά τα προσκόμματα της τόσο κατακαιρματισμένης ευρωπαϊκής αγοράς των 28. Συνάδελφοι από τον Μπερέκ δεν συμφωνούν διότι ισχυρίζονται ότι δεν χρειάζεται να επισκευάσουμε κάτι που λειτουργεί. Εγώ νομίζω πάλι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία και να ακολουθήσουμε μια άλλη ρότα. Κατόπιν, αξιολόγηση και follow-up του ε, ε, των κανονισμών. Θυμάστε, πρόκειται για μία απόφαση που πρέπει να λάβουμε σε σχέση με αυτούς που πρέπει να ταξιδέψουν στην Ευρώπη και τη χρήση των τοπικών δικτύων ε, κατά αντιδιαστολή με τους ε, εθνικού εθνικούς φορείς. Ε, αυτό μειώνει το κόστος. Οπότε θα πρέπει να εφαρμόσουν και αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας. Κατόπιν στις τηλεπικοινωνίες θα πρέπει να δούμε στα πλαίσια του 2020, συγγνώμη, 2020 ε, τι πρέπει να ε, αλλάξουμε πέρα από το να εξετάζουμε το ρόλο ε, του Μπέρεκ, τα γραφεία, την υποδομή, το προσωπικό, ε, ας έχουμε και μία ε, μελλοντοστραφή ευρωπαϊκή προοπτική. Σας ευχαριστώ συνάδελφε για όλες ε, τις, ε, συνάδε... για όλες τις παρατηρήσεις σας και για τις γεωγραφικού χαρακτήρα παρατηρήσεις σας και τις φιλοφρονίες σας και τα καλά λόγια για τη Ρήγα. Είναι όντως μια υπέροχη πόλη. Η κυρία Κωνσταντσε Κρέλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να συμπληρώσω λίγο και εγώ από πλευράς μου. Γεγονός, για πρώτη φορά πήγα εγώ στο Μπέρεκ και ε, χρειάστηκε να μάθω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το BEREC Office και το BEREC ε, σκέτο. Ε, το BEREC εκπροσωπεί τις εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και καλούνται να εφαρμόσουν αυτό που εμείς αποφασίζουμε ως νομοθεσία. Είναι γεγονός αυτό και πράγματι οι άνθρωποι κατασκοτώνονται και με μεγάλη επιτυχία. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, για μένα έχει σημασία να ασχοληθούμε με το δικό μας οργανισμό που είναι το BEREC Office που δεν είναι μόνο ο πιο πρόσφατος ευρωπαϊκός οργανισμός αλλά και ο μικρότερος και αν δω τι κάνουν εκεί υποστηρίζουν μεν το BEREC αλλά κανονικά θα πρέπει να υποστηρίζουν και τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αμέσως μετά την ίδρυση και ε, τη τα εγγένεια του BEREC Office ε, πέσανε οι περικοπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να κόψουν προσωπικό. Αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Και ε, σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε ε, στην ψηφιακή αγορά ε, θα έχουμε πολύ περισσότερη δουλειά, τεράστιο φόρτο εργασίας και ε, χρειαζόμαστε πολύ καλή ενημέρωση, τεκμηριωμένη και είναι ο ιδεώδης οργανισμός εκεί το BEREC Office για να μας υποστηρίζει ε, στη δουλειά μας. Και γι' αυτό Ε, για το επόμενο έτος ε, στις διαπραγματεύσεις του προϋπολογισμού καλό θα ήταν να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε περισσότερα χρήματα και περισσότερο προσωπικό για τον ΠΕΡΕΚ και με τη δική μας Επιτροπή Ήτρε να εκπονήσουμε μια στρατηγική για το πώς μπορούμε καλύτερα να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας έρχονται από εκεί και να ολοκληρώσουμε, να τα εντάξουμε αυτά περισσότερο στη δική μας δουλειά. Ελπίζω να συμφωνεί ε, ο κύριος Χέρπερ και με αυτά που λέω εγώ που συμφωνώ και εγώ με αυτά που είπε εκείνο προηγουμένω. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε. Και τρίτος, ε, που ήταν και εκείνο μέλος, ο κύριος Κρίστιαν Σκάρινς, που εκπροσωπούσε φυσικά και την Επιτροπή Ήτρε, αλλά και τη Λετωνική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη επίσκεψή μου στο Berek Office και πρέπει να σας πω ότι πάντα κανείς μαθαίνει κάτι παραπάνω. Θα συμφωνήσω και θα υποστηρίξω αυτά που είπαν οι δύο προλαλήσαντε συνάδελφοι. Μη λησμονείτε ότι το Μπέρεκ και το Μπέρεκ Office είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το Μπέρεκ είναι α πούμε εκεί που συνεδριάζουν οι εθνικοί ρυθμιστέ, ε, αλλά υπάρχει και το Μπέρεκ Office που είναι η υπηρεσία στη Ρήγα που είναι πάρα πολύ μικρή. Νομίζω ότι οι αριθμοί 17, 15 υπαλλήλου είναι η μικρότερη ε, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλάζει πάρα πολύ ε, συχνά με μεγάλη ταχύτητα το ε, προσωπικό. Ε, εκπλαγήκαμε όταν είδαμε ότι σε μια χώρα όπως η Λετωνία ε, έχουν δυσκολία να ε, πάρουν, ε, να, να προσλάβουν κόσμο, έρχονται όταν έρχονται εκεί, αλλά βλέπουν ότι στην ουσία πληρώνονται και πολύ λιγότερο γιατί υπάρχει ένας αλγόριθμος ένα συντελεστή ε, ο οποίο βασίζεται ε, στου μισθού τη της ε, και επομένω τελικά πληρώνονται τη τάξη του 0,75% πληρώνονται λιγότερο λοιπόν και φεύγουν πολύ γρήγορα. Είναι δύσκολο να κρατήσει κανεί το, ε, ε, τους υπαλλήλους ε, και σκέφτομαι ότι αν αυτό συμβαίνει σε αυτόν τον οργανισμό που, είναι στη, που έχει έδρα στη δικιά μου χώρα φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις νέων υπηρεσιών ή οργανισμών στο, σε άλλες χώρες. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε λίγο την ευρωπαϊκή διάσταση και όχι την ε, διάσταση την εθνική της χώρας γιατί διαφορετικά χάνουμε αυτήν την ευρωπαϊκή ε, ε, διάσταση. Εάν οι άνθρωποι αυτοί πληρώνονται καλύτερα, δουλεύουν καλύτερα και για μας. Ωραία, ωραία λέει ο Πρόεδρος. Εξάγουμε λοιπόν ήδη κάποια συμπεράσματα από την συζήτηση επόμενος ομιλητής, ιδιαίτερη περίπτωση σήμερα, ο Πολ Ρούμπιχ. Γιατί είναι η, η μέρα των γενεθλίων του, άρα είναι ιδιαίτερη μέρα. And uh, you know, colleagues, uh, Ξέρω ακριβώς πόσο νέος είναι, ξέρω ακριβώς τα χρόνια του, είναι νέος κυρίως συγκρινόμενος με μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει χρόνια πολλά και έχει το λόγο. Και για σήμερα το δωράκι σου είναι ότι δεν έχεις περιορισμό χρόνου ομιλίας. Ευχαριστώ πολύ. Το μεγαλύτερο δώρο προς τους συναδέλφους ε, είναι να μιλάω σύντομα και θα το τηρήσω. Ε, η συζήτηση για το Μπέρεκ είναι πολύ σημαντική. Εχθές είχαμε τη συνάντησή μας ε, και, την, ε, με την ΕΣΑ γιατί συνδέονται. Ε, είναι δύο δικοί μας τομείς αυτοί και έχουμε αγωνιστεί μαζικά να δημιουργηθούν. Και αν δούμε λοιπόν ότι υπάρχουν οι τεχνολογίες πληροφορίας, ε, τεχνολογίας ε, και συνδυάζεται με την ενέργεια διότι αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα και είναι και υποπίεση. Χρειάζονται περισσότερο προσωπικό. Το λέει και το ε, Μπέρεκ αλλά και ο Οργανισμός για την Ενέργεια και Ασφάλεια και θα ήταν να δούμε και τα δύο από κοινού γιατί Εμείς στην Ευρώπη ε, θα πρέπει ε, να προετοιμάσουμε την παροχή των συχνοτήτων τώρα, τις άδειε. Ε, και υπάρχουν κάποιοι κόμβοι στον ηλεκτρισμό που χρειάζονται ε, να τυποποιηθούν, να ε, γίνει μια συνεννόηση. Και αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, η ηλεκτρική ενέργεια λοιπόν και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Δεν ξέρω μήπως ε, θα ήταν καλό να συνδυαστούν, να συγχωνευτούν οι δύο οργανισμοί, διότι είδαμε και ότι στο περιαγωγή το roaming κυριαρχεί πολύ μεγάλος προστατευτισμός. Και το συγκεκριμένο θέμα τώρα το λύνει η αγορά. Το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο εθελοντικά έχουν καταργήσει ε, τα τέλη περιαγωγής. Και ε, υπάρχουν ε, κάποιες εταιρείες που αντιδρούν και η Google στο μεταξύ και στις τηλεπικοινωνίες ε, με τη νέα συσκευή και διαπραγματεύεται με πάνω από 100 εταιρείες τηλεπικοινωνιών και θα καταργήσει τα τέλη της περιαγωγής πολύ νωρίτερα από αυτό που δεν καταφέραμε εμείς να κάνουμε γιατί μπλοκάρουν τα κράτη-μέλη με τη δική μας νομοθεσία. Βλέπετε ένα παράδειγμα ε, και είναι το καλύτερο δώρο για νεθλίων μου αυτό. Η αγορά ρυθμίζει πιο γρήγορα από την νομοθεσία ένα ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας και όλους εσάς που πήγατε στη Ρήγα. Ε, στην αποστολή αυτή εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Ωραία. Και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη που είναι το υπαριθμόν 7 ε, για μια ευρωπαϊκή βιώσιμη βιομηχανία που να βασίζεται στα μέταλλα. Ε, ο εισηγητής είναι ο κύριος Ντουάχ Μαχτά, ο οποίος έχει προετοιμάσει και παρουσιάσει ένα έγγραφο εργασίας ε, που θα το συζητήσουμε. Έχουμε προβλέψει 45 λεπτά για την ανάπτυξη της βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας κοινών μετάλλων. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παρτέ για να μας παρουσιάσει τις απόψεις του για 5 λεπτά και μετά οι συντονιστές τρία λεπτά και τα ενδιαφερόμενα λοιπά μέλη δύο λεπτά έκαστος. Έχει το λόγο κύριε Μαχτά. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έλεγα μήπως ε, και μένα μου δίνατε ανοιχτό χρόνο ομιλίας, αλλά βλέπω ότι με περιορίζετε και επομένως θα περιοριστώ στα πέντε λεπτά. Πριν ε, ε, ξεκινήσω θα ήθελα να καλωσορίσω την παρουσία εδώ στην αίθουσά μας εργαζόμενους του εργοστασίου του Τάραντα από την Ιταλία και θα ήθελα να τους καλωσορίσω εξ ονόματος όλων. Είπατε πολύ σωστά ότι πρόκειται για μια ενδιάμεση άμεση παρουσίαση και όχι έκθεση. Ε, σκοπός της και πρόθεσή της είναι να ξεκινήσει την ε, ε, συζήτηση η οποία θα χρησιμοποιηθεί στο, στην έκθεση η οποία θα είναι ολοκληρωμένη περί τα τέλη Μαΐου. Θα ήθελα να σας εκθέσω τη μεθοδολογία εργασίας που αποφασίσαμε. Εμείς αποφασίσαμε να μιλήσουμε με τους βασικούς παραγωγούς των βασικών μετάλλων. Ήρθαμε σε επαφή με εκπροσώπους διαφόρων χωρών έτσι ώστε να συζητήσουμε και να συνδιαλλαγούμε μαζί τους, έτσι ώστε να δούμε τα σημεία απόκλησης αλλά κυρίως τα σημεία σύγκλησης και υπάρχουν ευτυχώς τέτοια. Πρώτον, όλοι συμφωνούν ότι πρόκειται για στρατηγικό τομέα για την Ευρώπη. Επίσης, όλοι συμφωνούν ότι ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Επίσης υπάρχει η θέση όσον αφορά τις αρμοδιότητες της τεχνογνωσίας και της ανάγκης να διατηρηθεί η τεχνογνωσία και να μεταβιβαστεί η τεχνογνωσία αυτή. Ε, υπάρχει επίσης ένα ζήτημα όσον αφορά την απόδοση των ποσοστώσεων και την κατανομή τους, ε, ένα πρόβλημα όσον αφορά την τιμή της ενέργειας και ένα άλλο ζήτημα τι σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση η αρμόδια αγορά θα τα αναπτύξω όλα αυτά εν συντομία. Διαπιστώσαμε επίσης ε, ότι όσον αφορά ε, τα μέταλλα της βασικής βιομηχανίας ε, να θυμίσω ότι είναι τα μη σιδηρούχα, είναι, είναι ο, ο και τα ιδιαίτερα μείγματα άνθρακα, ιδιαίτερες προσμίξεις τους. Αναφερόμαστε επίσης σε όλες τις εξορίξεις, εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς χαρακτήρα. Αναφερόμαστε τώρα σε ε, παραγωγές οι οποίες οπωσδήποτε είναι ενεργοβόρες, είναι ενεργοεντατικές και ε, δημιουργούν διοξίδιο του άνθρακα. Όμως ε, αυτό που είναι σημαντικό για τα μέταλλα είναι το ανταγωνιστικό στοιχείο που αφορά την τιμή. Αυτό που χαρακτηρίζει τον ανταγωνισμό τώρα είναι η καθαρότητα του μετάλλου και η τιμή του μετάλλου. Δεν είναι ένας τόνος ατσάλι, δεν είναι ίδιος με έναν άλλο τόνο ατσάλι. Ο χάλιβας δηλαδή ε, παρουσιάζει ιδιαίτερα ε, χαρακτηριστικά. Μιλάμε επίσης ε, για εργαζόμενους και για τεχνίτες με ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Να πω εδώ ότι η Ευρώπη έχει κλείσει πολλές εγκαταστάσεις. Έχουμε χάσει 60.000 άμεσες και 100.000 έμεσες θέσεις εργασίας σε μερικά χρόνια. Έχουμε με ε, περιπτώσεις ε, όπου κλείνουν εγκαταστάσεις ε, αλλά όπου οι ενδιαφερόμενοι μας λένε ότι εάν υπάρχει μια σχετική ανάκαμψη ενδεχομένως ένα-δύο χρόνια θα μπορέσουν να ξαναανοίξουν αυτές οι εγκαταστάσεις αλλά ότι σιγά σιγά κάποια στιγμή θα είναι δύσκολο έως αδύνατο να ξανανοίξουν διότι εντωμεταξύ θα έχουμε χάσει την τεχνογνωσία και τις ικανότητες. Ωστόσο υπάρχουν παραδείγματα εξαιρετικά Όπω όπως είναι αυτό της Γερμανίας όπου εξακολουθεί να υπάρχει κατάρτιση και μαθητεία έτσι ώστε να συνεχίσουν οι τεχνίτες να μαθαίνουν αυτές τις τεχνικές. Ε, σας τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι διαπιστώνουμε τώρα ε, ποια θα μπορούσε να είναι τα καθοριστικά στοιχεία έτσι ώστε να κινητροδοτηθούν οι επενδύσεις αλλά ε, και για να πω ότι στην ουσία δεν είναι τόσο ε, σημαντικό το ε, πρόβλημα των, του κόστους της, της εργασίας αλλά κυρίως το κόστος για το περιβάλλον και το κόστος για την πολιτική ε, γενικότερα και για το κόστος της ενέργειας. Ε, κοιτάξτε, αν μιλάμε για το περιβάλλον δεν υπάρχει μονάχα το διοξίδιο του άνθρακος, υπάρχουν και σειρά διοξινών. Δύο δευτερόλεπτα, δεν βλέπω να έχω πολύ χρόνο, αλλά δύο δευτερόλεπτα ε, για να σας πω ε, ότι πήγαμε στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής χάλιβα στην Ευρώπη αλλά αντιμετωπίζουμε δραματική κατάσταση γιατί έχουμε ε, τους ε, ανθρώπους οι οποίοι θέλουν την απασχόληση έχουμε, ακούμε ένα σωρό λόγια για την διατήρηση των θέσεων εργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά η οικογένεια Ρίβα του συγκεκριμένου εργοστασίου αθέτησε όλες τις υποσχέσεις της. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε ε, και τους ε, ε, κατοίκους της γύρω περιοχής που έχουν υποφέρει και εξακολουθούν να υποφέρουν από προβλήματα υγείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τη μία πλευρά δημιουργούνται πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας από τη βιομηχανία αυτή, αλλά οι θέσεις εργασίας δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν υλοποιηθούν εις βάρος της υγείας των ανθρώπων ή των εργαζομένων. Ε, θα ήθελα επειδή δεν έχω χρόνο να προχωρήσω γρήγορα να σας πω ότι χρειάζεται ε, ακολούθηση της διεθνούς αγοράς. Υπενθυμίζω ότι οι ανταγωνιστές μας, ε, ο ανταγωνισμός μας ο κύριος έρχεται από την Κίνα και δεν είναι δυνατόν να αφήσει η Ευρώπη αυτήν την εξοκοινοτική αγορά και δεν αναφέρομαι μονάχα στο, στον χάλιβα, αναφέρομαι και στον ανοξίδωτο χάλιβα και σε κάποια άλλα τα οποία είναι πολύ, κάποια άλλα και άλλα κράματα τα οποία είναι ε, ιδιαίτερα ε, προσοδοφόρα και σημαντικά για την Ευρώπη. Τώρα, εάν θέλουμε να δώσουμε ε, δωρεάν ποσόστοση θα πρέπει να, διοξιδίου του άνθρακος θα πρέπει ο άλλος να είναι διατηθειμένος να την αγοράσει. Ε, ε, ε, ναι αλλά αν, δεν μου δώσετε το χρόνο δεν θα μπορέσω να πάω, δεν θα μπορέσω να πω τα ουσιώδη. Ακόμη δεν τα έχω πει είναι σημαντικό ο αγοραστής ε, του, του ε, ε, κινέζικου χάλιβα να είναι υποχρεωμένος να αγοράσει από την ευρωπαϊκή αγορά αυτό, αυτή τη διαφορά που προκύπτει από το γεγονός ότι ο Κινέζος δεν θα λάβει υπόψη του ούτε το περιβάλλον ούτε τους, τις διατάξεις τις προστατευτικές ενώ αντίστοιχα ο Ευρωπαίος Ευρωπαίος παραγωγός ε, θα έχει επιβαρύνει την παραγωγή του με όλες αυτές τις ε, δεσμεύσεις. Ε, και να μην λησμονούμε ότι η διαρροή άνθρακα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς δεν μπορούμε να το, να το παραβλέψουμε. Η διαρροή του άνθρακα ξεκινάει από εκεί. Θα σας ξαναδώσω το λόγο μετά, μετά. Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση. Σας παρακαλώ λοιπόν συντομεύετε και περιμένετε λίγα λεπτάκια. Μιλήσατε 8 λεπτά συνολικά, ε, παρά είναι. Σταλίνη. Ε, Σαλίνη, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ για, αυτή, για αυτό το πρώτο προσχέδιο ε, το οποίο εισάγει σαν πρώτο στοιχείο που, το οποίο συμμερίζομαι την στρατηγική έποψη ε, του μέλλοντος όσον αφορά την ε, βιομηχανία του Χάλιβα. Μιλάμε για στρατηγικές ανάπτυξη στην Ευρώπη και όχι μόνο ε, θέτοντας την ψηφιακή ατζέντα, το ψηφιακό θεματολόγιο ε, στην κορυφή των ε, θεμάτων μας. Αλλά βεβαίως εδώ σήμερα η σιδηρουργία αλλά και η βιομηχανία γενικά είναι απαραίτητη έτσι ώστε να στηριχθεί στα πόδια του το οικονομικό μας μοντέλο και η, οικονομικό μας, και η οικονομική μας δομή η οποία βασίζεται στην εργασία και την ιδιοκτησία ιδιοκτησία ε, και ε, το εργοστάσιο είτε είναι μικρό είτε μεσαίο είτε μεγάλων διαστάσεων αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό το σχήμα. Ο εισηγητής ε, κατόπιν επικεντρώνει την προσοχή του και θα το πει και αργότερα στην στρατηγική προβλέποντας και ενδεχομένως ένα ξεπέρασμα του συστήματος ανταλλαγής εμπορίας ρήπων του ETS. Κοιτάξτε, εγώ ε, διαπιστώνω ότι χτες διακριτικά ολοκληρώθηκε ο τριμερής διάλογος ε, για, το, για την ανταλλαγή ε, καθώς επίσης για την ανταλλαγή ρήπων καθώς επίσης και για την διαρροή και αποθήκευση άνθρακα. Θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα δυνατότητες και για ένα ενδεχόμενο ξεπέρασμα, υπέρβαση αυτού του συστήματος όπως αφήνει να εννοηθεί ε, και το ίδιο το προσχέδιο της έκθεσης. Συχνά οι Ευρωπαίοι ε, δείχνουν να ενδιαφέρονται πολύ και ορθώς για το περιβάλλον, αλλά ενδιαφέρονται υπερβολικά λίγο ε, για την παρουσία και τον ρόλο της βιομηχανίας στην οικονομία και την οικονομική ανάκαμψη. Αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Ο συνάδελφος Τοσενόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, πολύ τον εισηγητή για αυτό το πρώτο έγγραφο εργασίας. Είναι περίπλοκο το θέμα και περίπλοκη η κατάσταση και προσπαθούμε να την περιγράψουμε. Είναι η βιομηχανία ε, των κοινών μετάλλων που είναι τα μη ευγενή μέταλλα και εξ όσων ε, γνωρίζω είναι από τα λίγα υλικά και τις ε, λίγες πρώτες ύλε ε, με τα οποία ασχολούμαστε εμείς στην Επιτροπή μας. Εδώ έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τη μεταποίηση ε, των μετάλλων και για την χαλιβουργία. Αλλά χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα θέματα, διότι η μεταλλουργία είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος και ε, από αυτόν εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο οι θέσει εργασίας ε, στο συγκεκριμένο κλάδο, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι κλάδοι ε, που είναι οι κατασκευές, η αυτοκίνητο-βιομηχανία. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς χάλιβα δεν στέκουν κυριολεκτικά πολλά κτίρια. Δεν θα μπορούσαν καν να οικοδομηθούν. ή θα ήταν πολύ προβληματικό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες εδώ για αυτά τα θέματα που άπτονται πολλών κλάδων της οικονομίας για να δούμε αν ε, θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε με δασμούς ε, αυτή τη βιομηχανία. Δηλαδή να γίνεται η προσαρμογή στα σύνορα. Γιατί υπάρχει ένα περιβαλλοντικό κόστος το οποίο θα πρέπει να αντισταθμίζεται. Δεν ξέρω, νομίζω διοικητικά κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Χαίρομαι πάντως που το συζητάμε το θέμα. Επίσης, ε, συμφωνώ με τον συνάδελφο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δεν είμαι υπέρ του συστήματος εμπορίας εκπομπών ε, στη Χαλιβουργία. Φοβάμαι ότι είναι πολύ μεγάλη αδυναμία. Ε, δεν λύνονται τα προβλήματα, μάλλον περιπλέκονται εάν εφαρμοστεί το e Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα τώρα ε, της ευρωπαϊκής ε, μεταλλουργίας, δεν έχουμε πάρα πολλές λύσεις. Αυτό που χρειάζονται είναι επενδύσεις και τεχνολογίες. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή στην Ευρώπη να υπάρξει τέτοια πίεση ώστε να παράγουμε λιγότερο χάλιβα και λιγότερα μέταλλα. Δεν εννοώ μόνο τις εγκαταστάσεις και τις θέσεις εργασίας που χάνονται, αλλά και γι' αυτό. Ε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο οι θέσεις εργασίας. Θα λείψει ο χάλιβας ως πρώτη ύλη από άλλους κλάδους της οικονομίας και θα πρέπει να εισάγεται. Με μεγάλο κόστος. Την Ευρώπη δεν θα πρέπει να τη συγκρίνουμε πάντα με την Κίνα. Μπορούμε να τη συγκρίνουμε και με τις ΗΠΑ Πολιτείες όταν μιλάμε για κόστος παραγωγής. Ε, πάντως χαίρομαι που μας απασχολεί αυτό το θέμα και θα πρέπει πιο συχνά να μας απασχολεί. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που ξεπέρασα το χρόνο μου. Αντιπρόεδρος Πέτερσεν εξ ονόματος των Φιλελευθέρων. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορούσε να έρθει ε, η σκιώδηση συγγήτρια και θα ήθελα να μιλήσω εξ ονοματής της εμ Συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι για το χάλιβα είναι χαμηλή η προσφορά και είναι υψηλέ οι τιμέ τη ενέργεια. Χρειάζεται αναδιάρθρωση, μεγαλύτερε, περισσότερε επενδύσει για να μπορέσουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο και να προσαρμοστούμε στην πράσινη οικονομία. Και γι' αυτό η Ευρώπη χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική πολιτική για να είναι ανταγωνιστικότερε οι τιμέ και πιο γενοτόματα προϊόντα. Επίση, οι πολιτικέ μα ε, για το περιβάλλον και για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα θα πρέπει να είναι κινητήριος δύναμη για να επέλθουν οι απαιτούμενε ε, τεχνολογικές αλλαγές ε, στον τομέα. Ε, επίσης θα πρέπει να το θέσουμε το ζήτημα στο γενικότερο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης. Θα πρέπει να μερμνήσουμε το ώστε να δημιουργηθεί μια νέα αγορά και να βελτιωθεί η βιομηχανία των κοινών μετάλλων, κυρίως ω προς την τιμή της ενέργειας, την πράσινη οικονομία, τη μετάβαση και την καινοτομία. Η διεθνώς ανταγωνιστικές ενεργειακές τιμές και ο ενεργειακός εφοδιασμός είναι βασικοί παράγοντες για το μέλλον αυτής της βιομηχανίας. Επίσης, ο κλάδος των κοινών μετάλλων είναι ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο όχι μόνο σε ευρωπαϊκό. Χρειαζόμαστε ω εκ τούτου ισότιμου όρου ανταγωνισμού ε, σε παγκόσμιο επίπεδο ε, και αθέμητη, αθέμητος ανταγωνισμό όπως το dumping ε, θα πρέπει να καταπολεμηθούν. Χρειάζεται λοιπόν σφαιρική προσέγγιση καθώ και ευέλικτα εργαλεία ούτω ώστε να έχουμε πρόσβαση και στην αγορά τρίτων χωρών. Γενικότερα η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι αποτελεσματική για να εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι και να εξασφαλιστεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε τις μελλοντικές συσκέψεις για την επεξεργασία του κειμένου. Σας ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρε. Ο κύριος Σιλικιώτης από την ΚΟΕΤΑ. Να ακούγεστε. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο μικρόφωνο, κύριε Σιλικιώτη. Τώρα εντάξει, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, να πω ότι ε, η σκιώδης εισηγήτρια της ΓΚΟΕ, η Παλώμα δεν μπορούσε να παρευρεθεί και θα κάνω εγώ την τοποθέτηση στη θέση τη. Ε, ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον Έντουα Μάρτιν για την σημαντική και ενδιαφέρουσα έκθεση που ετοίμασε, η οποία θα καθορίσει τι πολιτικέ προτεραιότητε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η βιομηχανία των κοινών μετάλλων είναι ένα σημαντικό τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Συμμεριζόμαστε του προβληματισμού και τι απόψει του εισηγητή, ιδιαίτερα όσον αφορά την υγεία των εργαζομένων και τον γειτονικό πληθυσμό. Θεωρούμε ωστόσο ότι είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε στην έκθεση και άλλα θέματα τα οποία δεν αναφέρονται. Αρχικά είναι σημαντικό να τονίσουμε πώ πρέπει να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή παραγωγή των μετάλλων καθώ και η διατήρηση αλλά ακόμα και η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασία στον βιομηχανικό τομέα. Στέχον μα πρέπει να είναι η βιομηχανία κοινών μετάλλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να καλύπτει τι ανάγκε των λαών, συμβάλλοντα ταυτόχρονα στην ανάπτυξη τη οικονομία. Είναι σημαντικό όμω η ανάπτυξη τη βιομηχανία μετάλλων να μην περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένε γεωγραφικέ περιοχέ. Θα πρέπει να προωθηθούμε συγκεκριμένα μέτρα ώστε να υπάρξει μια ισόρροπη εκβιομηχανοποίηση που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη όλη τη Ευρώπη. Εξίσου σημαντικό είναι να τονιστεί στην έκθεση ότι πρέπει να επανακαθορίσουμε του κανονισμού τη ανταγωνιστικότητα, οι οποίοι όπω έχει αποδειχθεί στην πράξη λειτουργούν προ όφελο μονάχα των μονοπωλίων και των πολυεθνικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο όπω αποδεικνύεται δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει τη βασική βιομηχανία για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκε τη κοινωνία, αλλά κατά την άποψή μα να προωθήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα. Πέραν αυτό, υποστηρίζουμε πλήρω την εσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστου στι τιμέ των μετάλλων ειδικά όσον αφορά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα στι τιμέ των μετάλλων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν το μέτρο θα συμβάλλουμε στην προσπάθεια περιορισμού τη καταστροφή του περιβάλλοντο, αλλά ταυτόχρονα θα προωθήσουμε και τα μέταλλα τη δική μα ε, εχώρια ε, παραγωγή. Εάν προωθήσουμε την άπτυξη τη βιομηχανία μετάλλων έχοντα ω νόμονα τι ανάγκε τη κοινωνία, ε, και τον εργαζομένο, τότε θα μπορέσει να συμβάλλει καθοριστικά κατά την μα στην άπτυξη τη οικονομία τη Ένωση, αλλά και στη βελτίωση τη ποιότητα ζωή των ανθρώπων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Oh, ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Από την FTD τώρα, ο συνάδελφος Μπορέλη, επίση συντονιστής, ή αντικαθιστά το συντονιστή. Α, όχι, είστε, είστε και ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα τον ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, για, το έγγραφο εργασίας το οποίο μας έστειλε τις προηγούμενες ημέρες. Θεωρώ ότι είναι απολύτως ε, θετικό να γίνει αναφορά ε, στην τροποποίηση, την αλλίωση της εσωτερικής αγοράς. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες, από τα μεγάλα μας στοιχεία προβληματισμού. Η βιομηχανία των κοινών μετάλλων ε, πρέπει να ανακάμψει στην Ευρώπη. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ανισορροπίες οι οποίες προκαλούνται από τις διαφορετικές φορολογικές πολιτικές ε, καθώς επίσης και από τη διαφορά του ενεργειακού κόστου στις χώρες μέλη. Υπάρχουν ε, οι οποίες έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ από την κρίση και επομένως αυτές θα έχουν πάντα μεγαλύτερο πρόβλημα και άρα το, η απόσταση που θα πρέπει να διανύσουν θα είναι πάντοτε μεγαλύτερη. Ένα άλλο στοιχείο είναι οπωσδήποτε η προσαρμογή των συνόρων. Ιδιαιτέρως κατά τη δική μου άποψη είναι ουσιώδους σημασία για τις εισαγωγές να εφαρμόζονται πάντοτε οι ίδιοι κανόνες όσον αφορά ε, το διοξίδιο του άνθρακα, ε, οι ίδιοι δηλαδή περιορισμοί που επιβάλλονται στους ενωσιακούς παραγωγούς, γιατί διαφορετικά θα υπάρχει πάντα πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους Ευρωπαίους και τους μη Ευρωπαίους παραγωγούς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Ε, τελειώσαμε του εκπροσώπου ε, των πολιτικών ομάδων και Καστήλιο Βέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Εδωά Μαχτά, γιατί έκανε ένα πολύ καλό έγγραφο εργασία και πάρα πολύ εύστοχο, πληρέστατο, ακριβέστατο, συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που πλήττουν ε, τη βιομηχανία κυρίως χάλιβα και αλουμινίου και τελικά όλη η βιομηχανική ενίσχυση της Ευρώπης βασίζεται σε δύο στοιχεία. Το ένα είναι η ανάπτυξη τεχνολογική που αυτό τον καιρό είναι η ψηφιακή κυρίως ανάπτυξη και αφορά και την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους κλάδους και η άλλη διάσταση είναι η ανάπτυξη των πρώτων υλών, έτσι δεν είναι, και των στοιχείων εκείνων που αποτελούν τη βάση για να μπορέσουν να δουλεύουν αυτές οι βιομηχανίες. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι αλληλένδετα και θα πρέπει να αναφέρονται από κοινού. Επίσης, είπε και ποια είναι τα βασικά προβλήματα της Ευρώπης αυτό τον καιρό το κόστος της ενέργειας και τα συμπαραμαρτούντα που συνδέονται με το κόστος για τις εκπομπές ρήπων. Δεύτερον, τα προβλήματα του εξωτερικού ανταγωνισμού που έχει η ευρωπαϊκή βιομηχανία ε, των μετάλλων και προτείνει ο εισηγητής να το συζητήσουμε και αυτό. Ε, ίσως να υπάρχει μια προσαρμογή στα σύνορα, γιατί όχι. Ε, είναι ενδιαφέρον να το συζητήσουμε, με τι άλλο. Μου άρεσε αυτή η σκέψη του. Και ένα άλλο στοιχείο που δεν συζητάμε ποτέ είναι τι γίνεται με τον ανταγωνισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και εκεί ζητήματα με ποιους όρους γίνεται ο ανταγωνισμός στην Ένωση. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή να κοιτάμε και προς τα έξω, αλλά να κοιτάμε και προς τα μέσα. Γιατί και εκεί υπάρχουν διάφορα εμπόδια. Λοιπόν, καλωσορίζω την πρόταση. Θα έχουμε το χρόνο μας να το συζητήσουμε με την ησυχία μας και σε λεπτομέρειες. Τίποτα άλλο και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Και τώρα, σκιώδης από τους πράσινους. Άρτια φιχθής, Ζαντό. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, ήμουν σε μια άλλη επιτροπή. Παρακολούθησα όμως... Ε, εκ του σύνεγγυς ε, την εργασία του συγητή και θα ήθελα να ε, χαιρετήσω την προσήλωσή του. Είναι απίστευτη αφοσίωση που δείχνει. Ε, μετήχα εξάλλου σε μία από τις αποστολές που διοργάνωσε και πραγματικά βρίσκω πως ε, για τα επιμέρους στοιχεία του φακελού είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να αντιδιαστέλουμε ε, τις παρατηρήσεις ε, που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο κοινοβουλίου, με τα σχόλια το, της βιομηχανίας, ε, των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών, των ενώσεων, των εργαζομένων, των μισθωτών. Και ξέρετε, γιατί ήσασταν και στην προηγούμενη θητεία, ότι αντίστοιχη δουλειά έχει γίνει για τη σιδηρουργία ε, είναι δουλειά, για τη χαλιβουργία, συγγνώμη, ε, είναι δουλειά ε, ουσίας και πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να τονίσω δύο βασικά ε, σημεία ε, της έκθεσης. Ένα δύσκολο ζήτημα καταρχάς για το Κοινοβούλιο που σχετίζεται εν μέρη με το ETS ε, την, ε, για τα ε, την εκπομπή ρήπων, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τη διαρροή άνθρακα. Πώς μπορούμε να επιβάλλουμε μέτρα στις βιομηχανίες μας όταν τίθεται εν κινδύνο η ίδια τους η ανταγωνιστικότητα και όταν αυτοί που δεν κάνουν καμία προσπάθεια τελικά γίνονται πιο ανταγωνιστικοί, μακροπρόθεσμα και πιο βιώσιμοι ε, σε σχέση με αυτούς που ε, καταβάλουν τις απαιτούμενε προσπάθειες. Πιστεύω ότι είναι σωστή η κατεύθυνση που ακολουθεί για αυτό το θέμα ο εισηγητή. Δεύτερο θέμα, το μεγάλο διακύβευμα ε, της, μελλοντική ανταγωνιστικότητα μελλοντικής ανταγωνιστικότητας Ξέρουμε ότι ε, υπάρχει βούληση από του εμπλεκόμενου φορείς ε, για τυποποίηση σε παγκόσμια κλίμακα ως προς τα κοινωνικο-οικονομικά πρότυπα, αλλά σίγουρα δεν μπορεί η ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη να βασιστεί σε μια κούρσα προς τα κάτω ε, η ανταγωνιστικότητά μας ε, θα πρέπει να ε, δράζεται σε αποτελεσματική χρήση των πόρων, σε ορθολογική χρήση των πόρων, σε περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, Είναι εξαιρετικά ποιοτική προσέγγιση του εισηγητή και ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εξαιρετικό έργο που έχει κάνει. Σας ευχαριστούμε κύριε Ζαντό. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Μαρτάν για την ε, έκθεση την οποία μας παρουσίασε. Ε, τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και χθες στην Επιτροπή Αναφορών με αφορμή καταγγελίες για τη λειτουργία του εργοστασίου του Τάραντα και χαιρετίζουμε την ευκαιρία αυτή την παρουσία των εργαζομένων ε, του Τάραντα, του εργοστασίου αυτού που είναι εδώ. Να πω λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι η μισθή ε, αλλά κυρίως ε, είναι, ε, όπως είπε και ο εισηγητής, η ποιότητα του μετάλλου, το κόστος της ενέργειας και οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν. Και νομίζω στο θέμα αυτό πλέον πρέπει να επικεντρωθούμε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για μια πολύ σημαντική βιομηχανία στην Ελλάδα που είναι η Λάρκο, η οποία είναι στις πέντε μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκόσμια που παράγει σίδηρο νικέλιο. Η ποιότητα του νικελίου είναι από τις καλύτερες στον κόσμο και όμως αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Και αυτό διότι έχει ένα κόστος ενέργειας 68 ευρώ την μεγαβατόρα, την ώρα που το, μέσος, το μέσο κόστος στην Ευρώπη είναι 25 ευρώ. Άρα λοιπόν το θέμα είναι τι επενδύσεις θα γίνουν γύρω από τα θέματα της ενέργειας, όπως επίσης και ε, γενικότερα τι παραγωγικές επενδύσεις για να μπορέσει να σταθεί αυτή η βιομηχανία. Επίσης ε, αντιμετωπίζουν τεράστια πρόβλημα και οι ελληνικές χαλιβουργίες με χιλιάδες θέσεις εργασίας πλέον να απειλούνται. Ε, φαίνεται ότι στην Ελλάδα τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά διότι και με τα μέτρα λιτότητας που έχουν ληφθεί οι βιομηχανίες, οι χαλιβουργίες έχουν χάσει πλέον το 85% των προϊόντων που μπορούσαν να παράγουν έχουν τεράστιες ζημίες. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να έχουμε μια διαφορετική στροφή στο ζήτημα της ε, στήριξης ε, των ε, βιομηχανιών των κοινών μετάλλων, να επενδύσουμε στην ίδια την παραγωγή, να επενδύσουμε πραγματικά στη βιομηχανία και να μην θεωρούμε ότι ο ανταγωνισμός με την Κίνα μπορεί να γίνει με την κινεζοποίηση των μισθών. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Επομένως, την ώρα που ο κύριος Δράγκη διαθέτει 1,13 ευρώ ουσιαστικά για την οικονομία καζίνο, εμείς θα πρέπει να διαθέσουμε τεράστια κεφάλαια στην ίδια την παραγωγή, στην ίδια την πραγματική οικονομία. Με αυτές τις κατευθύνσεις και τις παρατηρήσεις βεβαίως που έχει κάνει ο εισηγητής, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μέλλον για την βιομηχανία κοινών μετάλλων σε όλη την Ευρώπη και να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως είναι στην περίπτωση της Λάρκο που δεν πρέπει να οδηγηθεί σε ένα ξεπούλημα που θέλει να επιβάλλει η Τρόικα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να στηριχθεί η παραγωγή στο Νότο για να μπορέσουμε, στον Ευρωπαϊκό Νότο, για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να δώσουμε δουλειέ και προοπτική στι χώρε που αντιμετωπίζουν τεράστια ανεργία, όπω είναι αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα. Ευχαριστώ. Thank you very much, colleague, for your remarks. Σας ευχαριστούμε, συνάδελφε, για τις παρατηρήσεις. Η Πατρίσια Τόγια, η πρόεδρος. Και εγώ θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να ε, αναφερθώ θετικά τις παρατηρήσεις του συναδέλφου Μαρτά. Νομίζω ότι αγγίζει ε, πολύ σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων δεν και το σημαντικό ζήτημα που είναι το κόστος της ενέργειας ε, που βεβαίως έχει μεγάλο βάρος επί του τελικού προϊόντος και βεβαίως ε, που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη χαλιβουργία ορισμένων χωρών αλλά γενικότερα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ε, η ανταγωνιστική ικανότητα της Ευρώπης απέναντι σε άλλους παραγωγούς. Σήμερα αναφερθήκαμε στην Κίνα, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Ε, αυτό είναι, λέω, ένα κεντρικό θέμα. Ε, και η πρόταση που κάνεις είναι, εν πάση περιπτώσει, μία νέα πρόταση. Λιγότερο καλή, περισσότερο καλή μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει, αλλά πάντως θα πρέπει να την μελετήσουμε σε βάθος. Ο Μαρτάν λέει επίσης ε, ότι υπάρχει και το πρόβλημα της τρέβλωσης του ανταγωνισμού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω πάντως ότι βράχει πρόθεσμα και εν αναμονή ε, λύσεως πιο ε, σωστής με τους σημαντικούς παραγωγούς του, του κόσμου σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα των εσωτερικών ε, διαφορών. Ε, βλέπουμε ότι η Ιταλία, η Γερμανία δεν ε, βρίσκονται στο ίδιο, η Γαλλία δεν βρίσκονται ακριβώς στην ίδια βάση και το, το βάρος αυτού του προβλήματος γίνεται σιγά σιγά αβάσταχτο και επομένως θα πρέπει να βρεθεί ενδιάμεσα κάποια λύση. Δύο παρατηρήσεις για θέματα τα οποία θα πρέπει περαιτέρω να αναπτυχθούν ενδεχομένως μέσω των τροπολογιών. Το θέμα της έρευνας. Εδώ γίνεται αποδεκτό. Υπάρχει ήδη ε, ειδικό κονδύλι ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την έρευνα. Γίνονται λοιπόν εργασίες οι οποίες ε, μερικές φορές ε, έχουν ε, καταλήξει και σε κάποια πιλωτικά προγράμματα έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούν να δοθούν λύσεις στα πράγματα. Ένα δεύτερο το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ είναι της κυκλικής οικονομίας. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μεγάλος βαθμός ανακύκλωσης προϊόντων, στοιχείων τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να μειωθεί η ανάγκη εισαγωγής βασικών προϊόντων. Αυτό το σύστημα της ε, ε, κυκλικής οικονομίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι θέλουν να μπουν ε, σε αυτόν τον κύκλο αλλά δεν μπορούν γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τη βοήθεια η οποία ενδεχομένως μπορεί να παραχθεί ε, να παρασχεθεί συγγνώμη, ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο ε, αναφέρθηκαν από την Πιλάρ και από άλλους, δηλαδή θα πρέπει να ξαναδούμε οπωσδήποτε τους κανόνες του εσωτερικού ανταγωνισμού. Ο εισηγητής Εντουάρ Μαρτάν αναφέρεται στους κανόνες που θα πρέπει να ξαναδούμε όταν μιλάμε για συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε τους όρους όρους ε, της ε, ευρωπαϊκής ε, οικονομίας και του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να κάνει κάτι, να προχωρήσει λίγο όσον αφορά την αναθεώρηση των κανόνων του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να δούμε τα πράγματα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή, τον κύριο Μαρτάν. Δεν είναι ε, μόνο πολύ καλή η έκθεσή του, αλλά βλέπω για πρώτη φορά μια έκθεση με προτάσεις και όχι απλώς φωτογραφική καταγραφή μιας κατάστασης. Λαμβάνει υπόψη διάφορα στοιχεία ε, θα πρέπει να προσαρμοστούν διάφορα μέτρα που ισχύουν πέρα από τα σύνορά μας. Αυτό έχει να κάνει με την εσωτερική ανταγωνιστικότητα και απαντά και διάφορες ερωτήσεις ε, για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα. Ο κύριος Μαρτέν απαντά καταφατικά σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Επίσης, απαντά και διάφορα ερωτήματα που θέτουν εκείνοι που ανησυχούν για το περιβάλλον. Θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι όποιος θέλει να πουλήσει στην Ευρώπη θα πρέπει να φροντίσει να τηρούνται διάφορες προδιαγραφές και περιβαλλοντικές. Υπάρχει όμως εδώ ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Το διοξίδιο του άνθρακα το έχουμε λύσει εμείς στην Ευρώπη. Όχι βέβαια. Και σήμερα η Ανταρκτική ε, πλήττεται περισσότερο από όλα τα μέρη του κόσμου γιατί διευρύνεται η τρύπα του όζοντος. Έχει χαλιβουργία Ανταρκτική, όχι. Έχει άλλα εργοστάσια, όχι. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι που παράγουν χάλιβα αλλού ε, πρέπει να φροντίσουν να μειωθούν οι ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Το προτείνει ο εισηγητής. Λύση υπάρχει. Είναι εφικτή, είναι εφαρμόσιμη και με τις λύσεις αυτές που προτείνονται μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα εργασίας και προβλήματα ανταγωνιστικότητας και προβλήματα προστασίας του περιβάλλοντος και να τηρήσουμε και τους στόχους μας. Ελπίζω οι συνάδελφοι να υποστηρίξουν μαζικά αυτή ε, την αρχή για την προσαρμογή στα σύνορα. Ευχαριστώ. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη καινούργια γενική διεύθυνση αυτή. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ματία Πελεγκρίν, εξ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γαλλικά, μια και ο κύριος Μαρτά είναι, ε, είναι Γάλλος. Ε, πρέπει να πω ότι ε, ε, παλιότερα ε, ήταν ο κύριος Ματά και εκπρόσωπος εργαζομένων στην ομάδα υψηλού επίπεδου που είχε δημιουργήσει ο τότε αντιπρόεδρος Δαγιάννη. Ε, επομένως τον γνωρίζουμε πολύ καλά και γνωρίζουμε ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τον ε, τομέα και τη στρατηγική σημασία που έχει για την ε, Ευρώπη. Στο προσχέδιό του λέει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα γιατί όπως είπαν και οι βουλευτές οι οποίοι πήραν το λόγο αναφέρει θέματα τα οποία μπορούν να είναι και προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι προτάσεις και συστάσεις οι οποίες να αναφέρουν αναφέρονται μονάχα ε, στην Γενική ε, Διεύθυνση Γκρόαλα που είναι πολύ μεγάλη αλλά ε, και στην Πρίμα που είναι, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα θέματα αυτά οτιδήποτε σχετίζεται με την πρωτογενή αλλά και τη δευτερογενή παραγωγή όπως έλεγε η κυρία Τόγια προηγουμένως εντάσσονται στην ε, πολιτική της Κομισιόν. Επίσης στο πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 υπάρχει ένα τμήμα το οποίο αφορά και τις πρώτες ύλες και τα μέταλλα και είναι ένα τμήμα το οποίο διαχειρίζεται η δικιά μου μονάδα ε, και πρέπει να σας πω ότι χρηματοδοτούνται προγράμματα και στην πρωτογενή αλλά και στη δευτερογενή παραγωγή και συμμεριζόμαστε με αυτό που λέει η έκθεση ότι ε, δηλαδή βασιζόμαστε ε, στους τομείς του αλουμινίου και του άνθρακα θεωρώντας ότι είναι τομείς του μέλλοντος γιατί καμιά φορά αναφερόμαστε σε αυτά ε, τα θέματα λέγοντας ότι αυτά είναι τομείς του παρελθόντος όχι, είναι και τομείς του ε, μέλλοντος. Πρέπει να σας πω ότι ε, αποφασίστηκε από την Επίτροπο ε, η ομάδα υψηλού επίπεδου για τον Χάλιβα μετατράπηκε σε ομάδα υψηλού επίπεδου για την γενικότερη ε, βιομηχανική παραγωγή τέτοιων υλών. Η κυρία Κόσκα θα είναι η επικεφαλής και θα προεδρεύσει τις επόμενες συνεδρίασεις ε, και μετά τα θέματα θα προωθηθούν στο Συμβούλιο Βιομηχανίας. Ε, η ε, νέα Επίτροπος είναι αποφασισμένη να ακούσει την ισχυρή φωνή της βιομηχανίας γιατί υπάρχουν κοινά προβλήματα μεταξύ τους. Είναι τα προβλήματα του, του στρεβλωμένου δαθέμι του ανταγωνισμού, προβλήματα του ενεργειακού κόστους, ε, και βεβαίως ε, προβλήματα τα οποία προκύπτουν ε, από τους περιβαλλοντικούς κανόνες που έχουμε εμείς ενώ σε άλλες περιοχές του κόσμου δεν υπάρχουν. Η πρόταση που κάνει ο κύριος Μαρτάν όσον αφορά την προσαρμογή στα σύνορα, ξέρετε ότι είναι μία πρόταση ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη με την έννοια ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις επ' αυτού, αλλά βεβαίως θα συζητήσουμε και αυτή την ιδέα με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Κλίμα ε, που τώρα ε, βρίσκονται σε μία φάση σκέψης και τροποποίησης του συστήματος εμπορίας ρήπων ETS. Ε, επομένως όλα αυτά τα οποία εσείς προτείνετε θα μεταφερθούν στην DG Κλίμα και θα ληφθούν υπόψη όσον αφορά τις δόκιμες αγορές το έθιξε και η κυρία Τόγια προηγουμένως, ε, η ιστορία έδειξε ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αγορά ε, γιατί η αγορά του ανοξίδου του ε, ε, πρόκειται για μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Είδαμε και ότι ε, και στην περίπτωση του χάλιβα αλλά και στην περίπτωση του αλουμινίου και του ανοξίδου του ε, χάλιβα τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Είδαμε ότι είναι παγκοσμιοποιημένη αγορά με πολύ μεγάλες εισαγωγές από την Κίνα. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε και το θέμα αυτό. Thank Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρω πόσο σημαντικά όλα αυτά και τώρα ο συνάδελφος εισηγητής, όπως σας υποσχέθηκα άλλωστε κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο για δευτερολογία και πολύ χρόνο. Μέχρι και πέντε λεπτά δηλαδή αν επιθυμείτε για τα καταληκτικά σχόλια. Έχετε αρκετά θέματα να μιλάτε πέντε λεπτά. good. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε έχεις 15 λεπτά. Ε, γιατί εγώ είχα προβλέψει αρχικά να μιλήσω 15 λεπτά στην αρχική μου ε, παρουσίαση. Δεν μπόρεσα ε, να τα πω όλα αυτά που ήθελα, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε και τους άλλους συναδέλφους οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα και εμείς πρέπει να πω ότι προσπαθήσαμε να δούμε όσο γίνεται πιο γενικά το ζήτημα, να μελετήσουμε το μελετήσουμε από κάθε άποψη. Να σας πω λοιπόν ότι σας ευχαριστώ για τις ενθαρρύνσεις σας. Νομίζω πως όλοι κατάλαβαν πλέον ότι η αγορά των κοινών μετάλλων, των βασικών μετάλλων είναι κάτι ε, πολύ σημαντικό. Είναι μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και επομένως δεν μπορεί να μείνει ε, με ε, προκαταλήψεις και κλισές στο μυαλό της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, έγιναν κάποιες ε, ε, επικρίσεις ε, για την ε, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν και βεβαίως αυτό που είπε ο κ. Πελεγρίνης στο τέλος ότι δηλαδή είναι στρατηγικός ο ανοξίδωτος χάλιβας ναι είναι σημαντικό και βεβαίως το θέμα και του, των κραμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τελικά το έχουν και τις ανακύκλωσης ε, το έχουν ε, ε, πάρει στα χέρια τους κατά κάποιο τρόπο οι Κινέζοι και επομένως πρέπει να ανακάμψουμε όσον αφορά το τομέα αυτό. Ε, τώρα, η προσαρμογή στα σύνορα δεν είναι φόρος, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας βιομήχανος Ευρωπαίος να πρέπει να πληρώσει για να προστατέψει το περιβάλλον, πράγμα με το οποίο συμφωνούμε απολύτως, γιατί ένα πλανήτη τον έχουμε, άρα πρέπει να τον διατηρήσουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν ο Ευρωπαίος να πληρώνει έτσι ώστε να ε, ε, μπορέσει να ανταποκριθεί ανταποκριθεί στους ε, κανόνες ε, και μετά να εισάγονται προϊόντα ε, που έχουν παραχθεί με τελείως διαφορετικό τρόπο και διαφορετικό κόστος. Πρόκειται για ένα ποσό το οποίο θα βοηθήσει και την ευρωπαϊκή βιομηχανία και στόχος είναι στην ουσία η δημιουργία νέας υψικαμίνου και μάλιστα μιλούσαμε, μιλήσαμε με τους εμπλεκόμενους και ένας ε, ε, βιομηχα... βιομηχανός το, το πρόβλημα που έχει για να χτίσει μια καινούργια υψηκάμινο δεν είναι το κόστος το εργασιακό, είναι όλα τα υπόλοιπα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια παγκόσμια ε, διάσκεψη. Έξι δις ε, τόνοι είναι η κατανάλωση της Ευρώπης. Θέλουμε, ε, επομένως το ερώτημα είναι θέλουμε ακόμα μια τέτοια βιομηχανία στην Ευρώπη ε, και εγώ ε, προσυπογράφω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ότι δηλαδή η Κομισιόν στο πρόγραμμα που παρουσίασε την προηγούμενη χρονιά αναφέρει ότι θέλει την αναβίωση της βιομηχανίας, την, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, θέλει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να μεγαλώσει ε, στην Ισπανία ας πούμε έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, οι εγκαταστάσεις της Αλκοά δεν έχουν δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την, ε, τον ανταγωνισμό σε ένδο και έξω ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως αυτά θα πρέπει να τα δούμε στα πλαίσια της Ενεργειακής Ένωσης, να δούμε πώς είναι δυνατόν η Ευρώπη να επιτρέψει μακροχρόνια συμβάσεις. Οι Ισπανοί μας έλεγαν ότι πρέπει να ξέρουν για να κάνουν τον προγραμματισμό ε, πόσο θα κοστίζει ε, το, το μεγαβάτ ε, μετά από ένα χρόνο ή μετά από ενάμιση χρόνο. Ένα άλλο ζήτημα, το δόκιμο των αγορών, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και την ορατότητα που πρέπει να έχουμε. Ποια είναι όμως η ιδέα που έχει η Ευρώπη για τη βιομηχανία της. Ο κανόνας είναι να μην υπάρχει δεσπόζουσα θέση από μία χώρα ή από μία εταιρεία αλλά αν δούμε ας πούμε την περίπτωση της Κίνας και είναι η αλήθεια ότι δεν υπάρχει μόνο η Κίνα αλλά αναφέρομαι στην Κίνα γιατί ε, είναι ο κύριος ανταγωνιστής. Ε, βλέπουμε την πολιτική βούληση μιας χώρας να δεσπόσει επί της άλλης. Το βλέπουμε πίσω από τις, ε, ε, γιατί ε, διαπιστώνουμε ότι πίσω από τον ανοξίδωτο χάλιβα της Κίνας υπάρχει μια χώρα η οποία προωθεί την παραγωγή και την εμπορία. Αυτά όλα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ε, με την έκθεση αυτή και εδώ συμφωνούμε ε, με τους σκιώδεις ε, εισηγητές. Θέλουμε μία βιομηχανία ενωμένη, δυνατή, που θα σέβεται το περιβάλλον, που θα σέβεται τη δημόσια υγεία και ε, θα συμφωνήσω με αυτό που ο κύριος Ζαντού, αύριο οι επενδύσεις ε, στις ε, καθαρές μορφές ενέργειας, στη μείωση των εκπομπών ρήπων, στην σωστή ενεργειακή απόδοση, αυτά είναι θέματα τα οποία θα βοηθήσουν εν τέλει τη βιομηχανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε όχι μόνο για το έγγραφο, την έκθεσή σας, είναι καταπληκτικό, αλλά και για το πάθος που δείχνετε, το χρειαζόμαστε. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχετε ένα περιορισμένο αριθμό σελίδων για το σχέδιο έκθεσης, οπότε θα δυσκολευτείτε από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά έσω έτοιμος. 15-16 Ιουνίου του 2015 θα συζητήσουμε ε, το σχέδιο έκθεσης. Ε, τώρα θα περάσουμε στην ε, διαπραγματευτική εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό του 2016 Ανελή Μποσάουτ. Βαν Μποσάουτ, ζητώ συγγνώμη για την προφορά. Ε, δεν είναι τέλεια στα Ολλανδικά. Ε, είναι από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών η κυρία Μποσέιτ. Και ο στόχος, θυμίζω, για κάθε ε, γνωμοδότηση για την εντολή για το τριμερή διάλογο είναι να εξηγήσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες της Ήτρε. Το σημαντικότερο θέμα. Η κυρία Βανμποσάιτ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά, πολύ ωραία το είπατε το όνομά μου, Βαν Μποσάιτ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Πρόεδρε. Λάβατε το σχέδιο γνωμοδότησής μου ε, για τον προϋπολογισμό του 2016. Το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σχέδιο. Ε, είναι πολύ σφιχτές οι προθεσμίες υπήρξαν, γι' αυτό δεν ε, έχουμε το έγγραφο ακόμα σε όλες τις γλώσσες. Στην γνωμοδότησή μου προσπαθώ εγώ να εστιάσω στα ευρωπαϊκά θέματα προτεραιότητας. Είναι ένα προσχέδιο Ζητώ συγγνώμη, διακόπτει ο Πρόεδρος. Ε, παρακαλώ, οι ιδιωτικές συζητήσεις εκτός. Κυρία Τόια. Θα σας παρακαλούσα να καθίσετε ε, και τώρα θέλουμε να ακούσουμε την εισηγητριά μας. Παρακαλώ, κυρία Βανμποσόιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα Ολλανδικά έχει μια παροιμία που λέει «Οι απόντες έχουν πάντα άδικο». Οπότε συνεχίζω. Ε, είναι μια πρώτη πρόταση. Ε, περιμένω τις ε, τροπολογίες σας 21 Μαΐου έχει οριστεί από τη Γραμματεία η προθεσμία. Ε, να σας παρουσιάσω λίγο το έγγραφο. Το σημαντικότερο θέμα που θέλω να τονίσω είναι οι ε, περικοπές των ορίζοντα 2020 και η εξοικονόμηση από τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη για να χρηματοδοτηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Χρόνια ολόκληρα συζητάει το Κοινοβούλιο αυτά τα προγράμματα και είναι και άλλα προγράμματα που έχει πραγματικά προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή ε, ε, αυτή η προσπάθεια και δεν νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να χρηματοδοτήσει τα ίδια ρήξη και καινοτόμα προγράμματα. Αυτό το είδαμε και στα πρώτα προγράμματα που έπρεπε να εγκριθούν εντός εισαγωγικών από το ΕΦΣΥ. Ας είμαστε ε, σαφείς. Ε, θα πρέπει ορίζοντας 2020 και το συνδέοντας στην Ευρώπη να ε, διατηρηθούν όσοι έχουν. Δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από εκεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει πάρα πολύ εξονυχιστικό έλεγχο, όχι μόνο για αυτά τα θέματα, αλλά για όλες τις γραμμές του προπολογισμού. Υπάρχουν κάποια κακό κείμενα και αν τα διαπιστώνουμε είναι εξουσία μας να επεμβαίνουμε ως κοινοβόλιο. Έχουμε λάβει αυτή την εξουσία και θα πρέπει να την αξιοποιούμε. Προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ε, φέρει ξεχωριστή πρόταση για το 2016, τέλη Μαΐου θα μας φέρει, θα εξετάσω πραγματικά πολύ προσεκτικά και με κριτική ματιά ε, όλες αυτές τις γραμμές. Και πιστεύω και οι συνάδελφοι πρέπει να το κάνουν. Θέλω να πω το εξής, όταν ε, αναγνωρίζονται ε, κάποιες δαπάνες και δεσμεύονται κάποια λεφτά θα πρέπει να εκταμιεύονται. Ξέρετε ότι αυξάνονται τα ανεξόφλητα τιμολόγια χρόνο με το χρόνο και οι, οι μικρομεσαίοι δικαιούχοι ε, γνωρίζουν τεράστια προβλήματα από το γεγονός αυτό. Τα προγράμματα ε, είναι ε, πραγματικά διαφήμιση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εταίροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τα εκτελούν επί τόπου θα πρέπει και να πληρώνονται. Ε, ε, η γνωμοδότηση εστιάζει και σε θέματα προτεραιότητας για το 2016. Το ένα είναι το better ε, regulation θα πρέπει δηλαδή η νομοθεσία να είναι εφαρμόσιμη και ρεαλιστική και είναι από τα αγαπημένα μου θέματα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν ε, κάνει πολιτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει αυτή να αντανακλάται στα προγράμματα. Το πρώτο είναι η ενεργειακή απόδοση, το δεύτερο οι διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών και το τρίτο η κυκλική οικονομία. Ε, θα φροντίσω τα κονδύλια αυτά, οι γραμμές του προπολογισμού στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής να ε, τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. Αυτά θέλω να σας πω ότι είναι μια πρώτη μόνο πρόταση αυτή. Θα κάνω και άλλες ε, προτάσεις. Περιμένω τις τροπολογίες σας και ελπίζω να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς που να έχουν σου γίνεται ευρεία υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Μα, όντως, ε, θα πρέπει να παρουσιάσουμε τη δική μας γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ε, για ε, τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Το λόγο και ο κύριος Γκάιερ για να πει μερικά δικά του σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις από τη Σκοπιά ενός μέλους της Επιτροπής Προϋπολογισμών, που είναι και αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Παρατήρηση πρώτη αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Είναι προφανές ότι και ο προϋπολογισμός του 2016 θα έχει σημασία σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, διότι ε, θα πρέπει να χρηματοδοτήσει το Ταμείο Εγγυήσεων για αυτό, το Ταμείο Επενδύσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ επίμαχο στο Κοινοβούλιο για το πώς θα πρέπει να γίνει αυτό. Και ειδικά στην Επιτροπή μας και σωστά εκπροσωπείται η άποψη ότι θα πρέπει όσο γίνεται να προστατευτεί ο ορίζον 2020. Θα πρέπει όμως να έχουμε το εξής υπόψη μας σε αυτή τη συζήτηση με την απόφαση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ένα μεγάλο τμήμα των πόρων του προπολογισμού έχουν δεσμευτεί και είναι γνωστά. Δηλαδή κάθε κράτος μέλος γνωρίζει με μεγάλη σχετικά ακρίβεια τι ποσά ε, θα λάβει και τι ε, ποσά θα πρέπει να περιμένει από το Ταμείο συνοχή τα διευθυντικά ταμεία και τι πρέπει να εγγράψει στον προπολογισμό του από τη γεωργική πολιτική κτλ. Αυτό τι σημαίνει τώρα. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτό είναι λυπηρό, έχει πολύ λίγη και πολύ μικρή ελευθερία για μεταφορές πιστώσεων. Πήγαινε έλα εντός του προϋπολογισμού. Έχει πολύ μικρό περιθώριο λοιπόν στα χέρια της, αυτό που δεν είναι στους εθνικούς φακέλους, εθνικά κονδύλια, στα αγγλικά το λένε αυτό national envelopes και αυτό που δεν συνδέεται λοιπόν με τα κράτη είναι το ερευνητικό πρόγραμμα. Αυτό τι σημαίνει πάλι με τη σειρά του. Επιμένει το Κοινοβούλιο να κινητοποιηθούν από αλλού κονδύλια. Εάν γίνει κάτι τέτοιο θα ξανανοίξουμε το πακέτο του πολιετούς δημοσιονομικούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ε, δεινά ετών που θα μας βρουν και ε, θα έχουν τον τελικό λόγο τα κράτη-μέλη. Αυτό το αφήνω στην πολιτική φαντασία του ε, καθενός. Αν σας ενοχλώ να βγω από την αίθουσα, δεν έχω πρόβλημα. Τι έλεγα λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά μας εδώ. Δεν έχουμε πολλά λεφτά ελεύθερα με περιθώριο ελιγμών και έχει νόημα να κοιτάξουμε από ποιο ε, κονδύλι του προπολογισμού υπάρχουν χρήματα που μπορούμε να πάρουμε. Και τι να κάνουμε. Στον ορίζοντα 2020 αυτό συμβαίνει. Πού υπάρχουν μέσα και εργαλεία λοιπόν στον ορίζοντα 2020 που έτσι κι αλλιώς ε, είχαν ως στόχο να κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια για την έρευνα, όπως κάνει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Εκεί θα πρέπει βεβαίως να αποφύγουμε ε, δίπλη χρηματοδότηση, γιατί δεν θα υπήρχε και ε, προσθετικότητα. Ε, και μήπως στο πρόγραμμα αυτό το ερευνητικό έχουμε ήδη κάποιες δυνατότητες χρηματοδότησης και παράλληλα να κινητοποιηθούν λεφτά από το ΕΦΣΙ. Εκεί υπάρχει μια ευκαιρία να βρούμε χρήματα. Εγώ είμαι απολύτω στο πλευρό της Επιτροπής μας εδώ για την υποστήριξη και ε, ε, την προστασία του ορίζοντα 2000. Βεβαίως και χρειαζόμαστε θεμελιώδη έρευνα, ε, θέλουμε και έρευνα για την βιομηχανία, κοντά στη βιομηχανία, όλα αυτά είναι καλά. Αλλά να μην περιχαρακωθούμε σε μια θέση που να λέει δεν θα θυγούν τα λεφτά του ορίζοντα 2020. Γιατί έχω το μεγάλο φόβο ότι δεν μπορεί να σταθεί αυτή η θέση μας, ξέροντας και το συνολικό πλαίσιο. Εγώ θα το επιθυμούσα, αλλά οι εναλλακτικές λύσεις έχουν τεράστια περιπλοκότητα και τεράστια διάρκεια. Να πω τώρα και σε ένα δεύτερο θέμα που είναι οι διάφοροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Αυτό είναι ένα αντανακλαστικό θύμα. Όποιος γνωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω κάτω και ρωτήσει πού μπορεί να κάνει οικονομίες, το πρώτο θύμα είναι οι οργανισμοί. Βεβαίως έχουμε πολλούς και βεβαίως μόνο οι ειδικοί πρώτον μπορούν να απαριθμίσουν όλους τους οργανισμούς και μετά να πούνε και σωστά για ποιο λόγο υπάρχουν και τι σκοπό εξυπηρετούν, αλλά ε, αυτοί οι οργανισμοί ιδρύθηκαν ε, με πολύ καλή αιτιολόγηση και είχαν λόγο που έγιναν. Και τώρα υφίστανται τεράστια πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να κόψουν μόνο 5% στο προσωπικό, όπως λέει η Διοργανική Συμφωνία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις πιέζει, τους πιέζει πάρα πολύ να κάνουν και άλλες περικοπές ε, και μετατάξεις να βάλουν σε ένα πόλ τους υπαλλήλους για να μπορούν να τους ανταλλάσσουν. Ε, εγώ είμαι μόνιμος εισηγητής για τους οργανισμούς στην Επιτροπή ε, προπολογισμών που έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και μου έχουν γκρεμίσει τις πόρτες στο γραφείο οι οργανισμοί αυτοί με τις πιέσεις που ασκούν πάνω μου. Και ε, εγώ τους ενθαρρύνω, μιλήστε με τη μητρική σας επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόνο αυτή η Επιτροπή μπορεί ε, να αξιολογήσει με ακρίβεια το έργο το σημαντικό των οργανισμών, όπως είναι ο Μπέρεκ που αναφέραμε προηγουμένως. Και αυτό θα ήταν τεράστια βοήθεια και ανακούφιση για τους οργανισμούς αυτούς, εάν ακριβώς η γνωμοδότηση της αρμόδιας ε, επιτροπής τονίζει κάθε φορά ποια είναι η τεράστια σημασία του οργανισμού και πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και δεινή στην οποία έχει περιέλθει. Μόνο έτσι θα ασκήσουμε τεράστια πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει αυτό το, το redeployment pool. Εγώ μπορώ να βοηθήσω με τροπολογίες ήθελα να πω αυτά τα δύο είναι σημαντικά για μένα γιατί νομίζω και η πραγματογνωμοσύνη της Επιτροπής Ήτρε ε, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και στη δημοσιονομική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σα ε, Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Ε, είναι πολύ σημαντικές για μας. Χαιρόμαστε δε που εσείς ένα πλήρως ε, μέλος ε, της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Παρουσιάζεται και μια πολιτική άποψη σε σχέση με τις προτεραιότητες. Η... Τα σχόλια που κάνατε για τη χρηματοδότηση του ορίζοντα 2020 ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Τώρα από πλευρά τη Επιτροπή δεν είναι κανεί εδώ. Δεν είναι. Ό,τι κατάλαβα μπορούμε να στείλουμε το σχέδιο έκθεσης ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι, ούτως ή άλλως είναι υποχρεωσή μας αυτό. Θα του στείλω μια ενημερωτική επιστολή, γιατί είναι σημαντικό. Θα ήθελα και πάλι να πω πως η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες είναι στις 21 Μαΐου μέχρι τις 12 για τις ενδεικτικές προτάσεις για πιλωτικά προγράμματα. Η προθεσμία είναι στις 3 Ιουνίου, επίσης μέχρι τις 12. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση και πρέπει να αντιλάβουμε στα σοβαρά. Θέλει η συγγήτρια να κάνει κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις, παρακαλώ. Ναι, πολύ σύντομα. Είδα ότι ήταν και λίγες οι παρεμβάσεις. Ε, με εκπλήσει αυτό και μου κάνει εντύπωση οι σοσιαλιστές και δημοκράτες θέλουν να ανοίξουν την πόρτα για να μπει χέρι ε, στον ορίζοντα 2020 για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό για μένα είναι τελείως καινούριο. Πρώτη φορά τα ακούω και αυτά. Αγαπητοί συνάδελφοι. Οι τροπολογίες, νομίζω εγώ, είναι ένας πολύ καλός τρόπος ε, για να τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες επιτροπές. Ας περιμένουμε λοιπόν κάποιες εβδομάδες και τώρα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Όχι! Ναι! Δεν έχουμε άλλο σημείο για το πρωί. Σε τρεις ώρες. Στις τρεις το απόγευμα θα τα ξαναπούμε.